Good morning everybody. Ο πρόεδρος. Καλημέρα σε όλους. Κύριοι συμπρόεδροι, αγαπητοί φίλοι και βουλευτές, καλώς ήρθατε στις Βρυξέλλες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε σε αυτή την τόσο σημαντική εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ χαρμόσυνη έδειξη η σημερινή εκδήλωση αυτό το Ευρωπαϊκό Φόρουμ των Τόμων με ειδικέ ανάγκες και με την ευκαιρία να σας ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε και τώρα να μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα μπορείτε να μιλήσετε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες σήμερα εδώ. Η σημερινή εκδήλωση αφορά 80 εκατομμύρια συμπολιτών μας που έχουν ειδικές ανάγκες σε μόνιμη βάση αλλά υπάρχουν και άλλοι τόσοι που έχουν κάποια προσωρινή αναπηρία και αυτοί βέβαια αξίζουν της προσοχής μας θέλουμε να παράσουμε κάποιες εγγύσεις ότι υπάρχει η Ευρώπη των ευκαιριών της ελευθερίας και να είναι μια πραγματικότητα για όλους μας η ένταξη, ενσωμάτωση είναι θεμελιώδης ε, αξία. Έχουμε αυτό το κοινωνικό μας μοντέλο, το οποίο δεν είναι δυνατόν να αφήσει εκτός κανένα. σήμερα θα πρέπει μαζί να μια νέα όθηση αυτή την προσπάθεια. Το πρόβλημα της ε, αναπηρίας είναι προτεραιότητα στο θεματολογιό μας και πλευράς πολιτικής και κοινωνικής. Ανέκαθεν το κοινοβούλιο είναι μάχη για αυτή την υπόθεση, να ληφθούν μέτρα τόσο ώστε να υπάρχει πλήρη συμμετοχή στις εργασίες μας ε, σε ανθρώπους με αναπηρία. Είτε πρόκειται για το προσωπικό μας, τους συνεργάτες μας, είτε πρόκειται για βουλευτές. Οπότε και σήμερα θα πρέπει στην σημερινή συνάντηση πέραν των 23 ε, επισήμων γλωσσών μας να έχουμε ε, την νοηματική γλώσσα και τον Μπράιτ και την στενογραφία. Οπότε θα πρέπει να προσαρμοστούν όλα αυτά τα δούμε με αναπηρία στι εργασίε μας, αλλά κυρίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προσαρμοστεί στις ανάγκες των ανθρώπων αυτών. Είναι θέμα ελευθερίας. Θα πρέπει όλοι να μπορούν να εργαστούν, θα πρέπει να μπορούν να εκφραστούν στο Κοινοβούλιο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το πιο ολοκληρωμένο που προσυδειάζει την προσωπικότητά τους. Κατόπιν ε, έχουμε ιδιαίτερε ε, ρυθμίσεις για τους ε, ανθρώπους με απειρία και τα παιδιά τους. Και έχουμε κάποιες δομές οι οποίες είναι τέτοιες που προσαρμόζουν και το ακτήριο του Κοινοβουλίου όσον αφορά την προσβασιμότητα, όσον αφορά την ενσωμάτωση. Άρα θα πρέπει να υπάρξει εγγύθητη συμμετοχής των πολιτών παντού και όχι μόνο στις Βρυξέλλες αλλά και στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι απαράδεκτο να παραμένει εμπόδιο για να για όποιον θέλει να συμμετάσχει στο δημοκρατικό γίγνεσθε. Δυστυχώς όμως ε, ακόμα έχουμε πολλές χώρες της ε, Ένωσης που να κάνουν τέτοιε ενέργειε και μία από τις πρώτες μου πράξεις ω Προέδρου ήταν το να απευθύνω μία επιστολή σε όλους τους διαφορετικούς κρατών και κυβερνήσεων και τους ε, ζήτησα να παράσχουν εγγύηση σε όλους τους ε, πολίτες με την ευκαιρία των επερχομένων ε, ευρωπαϊκών εκλογών να τους παράσχουν την εγγύηση λίγο της ελεύθερης ψήφου και ιδιαίτερα να πλαισιώσουν τα άτομα με αναπηρία. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε με καμπάνιες πληροφόρησης στις οποίες όλοι έχουν πρόσβαση και έχουμε αυτό το μνημόνιο ε, προθέσεων όσον αφορά ε, την οργάνωση της ε, Μαδρίτης για τα άτομα με προβλήματα όρασης. Και είπαμε ότι αυτό θα πρέπει να επεκταθεί παντού όπου έχει γραφεία και εκπροσώπηση η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπότε και εσείς οι 700 εκπρόσωποι των σχετικών φορέων παρακαλώ να εκμεταλλευτείτε αυτή την ευκαιρία και θα πρέπει να δώσουμε σε όλους εγγύηση πλήρου συμμετοχής για κάθε τομέα απασχόλησης, παιδείας, δημόσιες υπηρεσίες, μεταφορές, πολιτιστικά, τουρισμό. Σίγουρα έχει σημαθεί πρόοδος ε, τα τελευταία χρόνια, αλλά μπορούμε και οφείλουμε να κάνουμε ακόμα πολλά περισσότερα. Η έκθεση όσον αφορά την πρόοδο ε, τη στρατηγικη 2010 2010-2020 της σχετικής στρατηγική που δημοσιοποιήθηκε τον Φεβρουάριο φέτος αναφέρει τις ε, πρόοδες που έχουμε σημειώσει μέχρι σήμερα και το τι θα πρέπει ακόμη να κάνουμε. Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να μας βοηθήσουν σημαντικά και ε, επίσης να υπάρχει πιο, πιο εύχριστα τα, τα διαδικτύου να μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση σε κάθε δημόσια διοικητική υπηρεσία και θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε και το δορυφορικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Γαλιλαίων. όσο ήμουν επίτροπος πρώτα μεταφορών και κατόπιν με το χαρτοφυλάκιο της βιομηχανίας, ε, τρέξαμε ένα πρόγραμμα περισσότερα από ένα προγράμματα είναι αλήθεια και αυτοί που είχαν προβλήματα κινητικότητας μπορούσαν με αυτό το πρόγραμμα να πλαισιωθούν, να μπορέσουν χωρίς βοήθεια να χρησιμοποιήσουν ε, αυτό το περιφορικό σύστημα και η προσπάθεια αυτή απέδωσε καρπούς και ποιήσεις, ε, υπάρχουν εφαρμογές δηλαδή μπορούν αυτοί που έχουν πρόβλημα όρασης να χρησιμοποιήσουν κάποια γυαλιά και κάποιο ακουστικό και έτσι επί τη βάση κάποιων οδηγιών, κάποιων σημάτων δορυφορικών ε, μπορούν αυτοί που έχουν μειωμένη όραση ή που ε, πάσχουν από τύφλωση να μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς να είναι υποχρεωμένοι, να έχουν κάποιο συνοδό ή κάποιο ζώο ή ε, έχουν τουλάχιστον αυτό το, το μπαστούνι Αυτά είναι σημαντικά βήματα προόδου και έχουμε τόσες εφαρμογές και κάποιες σύγχρονες εφαρμογές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε την, το πρόσφατο σχέδιο οδηγίας και έτσι προβλέπονται κάποιοι κανόνες ούτως ώστε ε, να μπορούν τα πρόσωπα που έχουν πρόβλημα όρασης να έχουν πρόσβαση σε πολιτιστικά έργα πέραν των δικαιωμάτων του δημιουργού και είπαμε είναι και θέματα μηδία αναγνώριση, και αυτά θα πρέπει να επεκταθούν σε όλα τα κράτη-μέλη. Ως ε, Επίτροπος Μεταφορών μπόρεσα να βοηθήσω για αυτό τον κανονισμό που διευκολύνει τα 130 εκατομμύρια των ανθρώπων με κινητικά προβλήματα να μπορούν ως επιβάτες να διακινηθούν στα αεροδρόμια με περισσότερη ευκολία, με συγκεκριμένες ρυθμίσεις, συγκεκριμένες διαδρομές και έτσι να ε, μπορούν όλοι να απολαύσουν την ελευθερία της διακίνησης. Και για μένα δεν ήταν θέμα μόνο αλληλεγγύης ήταν πάνω απ' όλα ένα θέμα ελευθερίας. Γιατί η λέξη ελευθερία είναι σύμβολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την χαρακτηρίζει, είναι η σημαία της, είναι θεμελιώδης αξία της. Πάνω ακόμα έχουμε πολλούς φραγμούς αρχιτεκτονικούς, οπότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν περιφερειακά ταμεία, ε, ταμείο επενδύσεων ε, μέσω του προπολογισμού μας. Και έτσι ε, μπορούν όλοι να ωφεληθούν από μια ευελιξία του προπολογισμού και στην ε, βιοιατρική, στη σχετική έρευνα, να βοηθήσουμε την κινητικότητα και να αξιοποιηθεί το πρόγραμμα Horizon 2020 και τα αντίστοιχα μέλλοντα προγράμματα να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτω ώστε αυτή η πρωτοπορία την οποία έχει η Ευρώπη να συνεχιστεί. Πρόκειται για κάποιε προσπάθειε ερευνητικέ, επιστημονικέ και έτσι να προσφέρουμε και απασχόληση ε, σε αυτά τα πρόσωπα δουλειά. Θα πει αξιοπρέπεια. Θα πει και αυτή η λέξη ελευθερία και θα πρέπει να υπάρχει τέτοιου είδου ε, κατανόηση εγγύηση ισότητα για όλου. Πάντω η ανεργία πάει στο 20%, 20% ε, κάτω από την ανεργία προσώπων που δεν έχουν κάποια αναπηρία. Και πέρσι το Κοινοβούλιο ε, προσπάθησε να υπάρχει ο ίδιος ορισμός της ε, αναπηρίας σε όλα τα κρατημέλη όσον αφορά τη λειτουργία της αγοράς εργασίας. Γιατί υπάρχουν διαφορές μεταξύ κρατών μελών και γι' αυτό και θέλουμε να υπάρχει ε, αντιστοιχεία και έτσι να μην γίνονται δεσμενείς διακρίσεις από πλευράς εργοδοσίας. Εναρμόνιση επομένω σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα πρέπει να εφαρμοστεί η οδηγία για την ισότητα μεταχείρισης και η σχετική σύμβαση του ΟΗΕ. Επομένως, δημιουργία απασχόλησης θα πει να γίνει κάτι στην πραγματική οικονομία και θα πρέπει το, το κράτος και ο ιδιωτικός τομέας να συνεργαστούν και έτσι τα πρόσφατα αναπηρίες να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και αυτό θα πρέπει να γίνει και με δημόσιες συμβάσεις. Ε, γνωρίζετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πρόκειται να εφησυχαστεί όσον αφορά την υπεράσπιση των συμφερόντων σας. Ευχαριστούμε την διακομματική ομάδα. Είναι από τις πιο παλιές μας διακομματικές ομάδες εδώ το Κοινοβούλιο γιατί πάντοτε είχαν σημαία τους στην υπεράσπιση των προσώπων με αναπηρία στο Κοινοβούλιο αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Και επίσης να ευχαριστήσω ιδιαίτερως τον συνάδελφο Μάρεκ για όλα όσα έκανε όσον αφορά την ένταξη, την ενσωμάτωση. Ένα χειροκρότημα για τον Μάρεκ Πλούρα με τις ευχαριστίες μας. Nel 2015 abbiamo... 15 φτιάχνει αυτό το δίκτυο βουλευτών. Πρόεδρος είναι ο συνάδελφος Άνταμ Κόζα, ώστε να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε την ε, συμφωνία του ΟΗΕ για τα πρόσωπα με αναπηρία. Και πάλι ευχαριστούμε Άνταμ αλλά και εσένα Μάρεκ. Αυτό το δίκτυο ε, καλύπτει εκπροσώπους των 12 νομιστών Επιτροπών, τόσο να υπάρχει κάποιο συντονισμό για την ε, δράση μα υπέρ αυτή τη σύμβαση. Και επίσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να ε, φτιάξει μια υπηρεσία όσον αφορά κάποια ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Επίσης, πανεπιστημιακό δίκτυο που θα διατυπώσει προτάσεις προς τα κράτη-μέλη. Και λόγω της πολύτιμης Συμβουλής της Elgar Stevens εγκρίναμε την περασμένη εβδομάδα αυτό το κείμενο, αυτό το ψήφισμα όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα πρόσωπα με αναπηρία. Ευχαριστώ για όλα όσα έχετε κάνει και εσείς. Είναι ξεκάθαρο ότι θέλουμε ότι το ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε τη στρατηγική μας και να την ενσωματώσουμε σε πάσα πολιτική της ε, Ένωσης στη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου υπάρχει ένας πάγιος διάλογος με όλους τους ώστε να ξεκαθαρίσουμε μια στρατηγική για μετά το 2020 που θα αφορά την αναπηρία. Και ξεκινούμε με την δική οργάνωση, το φόρουμ το δικό σας, διότι θα πρέπει καμία απόφαση να λαμβάνετε χωρίς εσείς να συμμετάσχετε. Ναι, καμία απόφαση στην Ευρώπη δεν πρέπει να υπάρχει χωρίς την γνώμη σας. Οπότε θα πρέπει να σου πω ότι οι πόρτε μας είναι πάντοτε ανοιχτέ για εσά για την συνεργασία μαζί σα. Και όχι μόνο για σήμερα που έχουμε αυτή την ευκαιρία, μια από τι πιο σπουδαίε εκδηλώσεις που έχουμε οργανώσει εδώ στο Κοινοβούλιο. Η πόρτα του Κοινοβουλίου πάντα είναι ανοιχτή, ούτω ώστε να φουγκραστεί τις προτάσεις σας, εσάς, και έτσι μαζί να χαράξουμε το μέλλον μας ε, ε, ημών των ε, Ευρωπαίων Ελευθέρων Πολιτών. Καλώς ορίσατε στις Βρυξέλλες. Ora la parola al Presidente del Forum Europeo delle Persone. Τώρα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ανθρωπίνων Περίοδο, ο κ. Βαρδακαστάνης έχει το λόγο. Αξιότιμη, αξιότιμη Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, αξιότιμοι ε, συμμετέχοντες, ε, μέλη, επισκέπτες, ευρωβουλευτές, συνάδελφοι από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Πρόεδρε, βρισκόμαστε εδώ από την Ανατολή και τη Δύση, το Βορρά και το Νότο. Η πολυμορφία της Ευρώπης είναι παρούσα στην αίθουσα. Θα ήθελα εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Αναπηρικού Κινήματος να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του συναδέρφους του, τις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε κατά τη διοργάνωση αυτής της πολύ σημαντικής εκδήλωσης. Όπως πολύ εύστοχα επισημάνατε κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη από την σύστασή του ήταν έθερμος υπέρμαχος και υποστηρικτής των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Και όντω η διακομματική ομάδα των ατόμων με αναπηρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι από τις ε, πιο παλιές και πιο δραστήριες διακομματικέ ομάδες για τα άτομα με αναπηρία. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμότατα όλα τα μέλη της διακομματική ομάδα για την προσήλωση, την αφοσίωση και την υποστήριξή του. Θα ήθελα επίση να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που βοήθησαν τις αντιπροσωπείες μας ε, για να μεταβούν στις Βρυξέλλες από τα κράτη-μέλη. Σήμερα έχουμε το τέταρτο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, για άτομα με αναπηρίαση. Η πρώτη εκδήλωση έγινε το 1993 για να εορτάσουμε την πρώτη Διεθνή ημέρα των ατόμων με αναπηρία, που ήταν η 3η Δεκεμβρίου. Το δεύτερο τέτοιο φόρουμ έλαβε χώρα στα τέλη του 2003, όταν ολοκληρώθηκε το πρώτο και μοναδικό έτος των ατόμων με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό, κύριε Πρόεδρε, απευθύναμε έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ζητήσαμε τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να ξεκινήσουμε μια νέα δεκαετία με ανανέωση αυτής της κινητοποίησης της κοινωνίας ε, των διαφόρων φορέων, των πολιτικών ηθινόντων και όσων λαμβάνουν αποφάσεις ε, για τα άτομα με αναπηρία, οργανώνοντας το δεύτερο ευρωπαϊκό έτος για τα άτομα με αναπηρία το 2021. Και είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι αυτές οι δύο εκδηλώσεις έλαβαν χώρα σε μια περίοδο επέκτασης, διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, η τρίτη τέτοια εκδήλωση έγινε το 2012 σε πολύ ταραχώδεις καιρούς, σε μια περίοδο οικονομικής, χρηματοπιστωτικής και για μερικές χώρες και κοινωνικής κρίσης. Και τα πρώτα θύματα αυτής της κρίσης ήταν και είναι τα άτομα με αναπηρία, με πολύ σημαντική οπισθοδρόμηση των δικαιωμάτων τους. Αυτή η τέταρτη εκδήλωση, αυτό το τέταρτο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των Ατόμων με Αναπηρία γίνεται σε μια περίοδο που την χαρακτηρίζουμε ως περίοδο ανάκαμψης. Χρειαζόμαστε λοιπόν τώρα μια νέα όθηση, μια νέα φόρα, μια νέα ορμή για να επανέλθουμε στις βασικές ζωτικές και θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί έχουμε πια τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, έχουμε τη Σύμβαση, έχουμε τα μέσα και τα εργαλεία. Χρειαζόμαστε λοιπόν μία ισχυρή συλλογική βούληση από όλα τα θεσμικά όργανα. Μία βούληση αντάξια με τη δική σας, με την βούληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και ελπίζω ότι θα καταφέρετε να συγκαλέσετε εδώ τη δεύτερη συνεδρίαση των τριών προέδρων, του κυρίου Γιουνκέρ, του κυρίου Τούσκ και του, του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η πρώτη τέτοια συζήτηση έγινε το 2011 για να συζητήσετε τις θεσμικές διοργανικές ρυθμίσεις που είναι απαραίτητες προκειμένου να μπουν τα θεμέλια για, τα, για τις ανάγκες μας της επόμενες δεκαετίες για τις οποίες θα μιλήσω αργότερα. Σε αυτή την βαρισίμαντη ε, εκδήλωση σήμερα, όπου θα εγκρίνουμε δύο πολύ σημαντικά έγγραφα. Το πρώτο αφορά την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στις ευρωεκλογέ του 2019. Πρόκειται για το μανιφέστο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία για τις επόμενες ευρωεκλογέ. Το δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεστε, τη συμμετοχή στον πολιτικό βίο. Αυτά είναι τα δύο δικαιώματα. Τα δικαιώματα του εκλέγην και του εκλέγεστε. Και ξέρουμε ότι εκατοντάδε χιλιάδες ε, άτομα με αναπηρία έχουν στερηθεί ε, των εκλογικών τους δικαιωμάτων. Και πραγματικά άκουσα με μεγάλη αγαλίαση τα λόγια σας και τα επιτεύγματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να γίνουν προσβάσιμες οι εκλογές και για τα άτομα με αναπηρία. Και αυτό ήταν πολύ ισχυρό το μήνυμα που θα πρέπει να, να σταλεί προς τα κράτη-μέλη και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να μεριμνήσουν και να άρουν τους φραγμούς και τα εμπόδια που εμποδίζουν τα άτομα με αναπηρία να ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα του πολίτη. Γιατί το ερώτημα είναι απλούστατο. Είμαστε πολίτε ή δεν είμαστε. Γιατί αν δεν έχουμε το δικαίωμα του εκλέγην, αν δεν έχουμε το δικαίωμα ψήφου, δεν είμαστε πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι ένα αίτημα, ένα πάδημο αίτημα που απευθύνουμε στους πολιτικούς ηθήνοντες σήμερα. Το δεύτερο έγγραφο που θα εγκρίνουμε είναι μια πολύ σημαντική πράξη, ένα πολύ σημαντικό ψήφισμα για τις για την επόμενη δεκαετία. Χρειαζόμαστε μία πανευρωπαϊκή στρατηγική για τα άτομα με αναπηρίες γενική, πλήρη, περιεκτική που θα καλύπτει τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία τις επόμενες δεκαετίες. Και επίσης θα πρέπει να κυρωθεί η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών. Η υπογραφή έγινε στα μέσα της κρίσης και θα ήθελα να πω ότι μέχρι στιγμής όλα όσα έγιναν είναι καλά, θετικά τα επιτεύγματα, μέχρι στιγμής όλα καλά, με μία εξαίρεση όμως κύριε Πρόεδρε. Τα κοινοτικά θεσμικά όργανα δεν ζήτησαν από τις χώρες ε, που εφάρμοζαν πολιτικές λιτότητες να προστατεύσουν περισσότερο τα άτομα με αναπηρία. Δεν τους το ζήτησαν. Και είναι υποχρέωση των κοινοτικών θεσμικών οργάνων να απευθύνει τέτοια απέτηση στα κράτη-μέλη. Και αν οι κυβερνήσει των χωρών αυτών ισχυρίζονται ότι τα κοινοτικά θεσμικά όργανα του ζήτησαν ε, να λάβουν μέτρα για να περικόψουν τα δικαιώματα και τα προνόμια των ε, ατόμων με αναπηρία, θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και τα ε, θεσμικά όργανα. Η νέα δεκαετία που θα ξεκινήσει με το δεύτερο ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με αναπηρία και μια εύρωστη και περιεκτική στρατηγική για τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να υιοθετήσει μια σφαιρική προσέγγιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και να επιστρέψουμε στις πραγματικές ρίζες των ευρωπαϊκών αξιών. Και φυσικά αυτή η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να είναι πλήρως ε, ενσωματωμένη στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν περάσει 20 χρόνια από την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Φόρουμ των Ατόμων με Αναπηρία. Οπότε σήμερα γιορτάζουμε και την 20 ετία της δράσης μας, της παρουσίας μας. Γιορτάζουμε τα 20 χρόνια της κινητοποίησής μας και της ε, επισήμανσης των προβλημάτων των ατόμων με αναπηρία στους πολιτικούς ηθήνοντες. Και όπως είπατε κύριε Πρόεδρε, το σύνθημά μας και η αρχή μας είναι τίποτα για μας χωρίς τη συμμετοχή μας. Και μάλιστα έξω από την αίθουσα έχουμε και μία έκθεση φωτογραφίας για την 20η αυτή ιστορία του Ευρωπαϊκού Φόρουμ των Ατόμων με Αναπηρία. Θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω θερμότητα, θερμότατα όλους τους συναδέλφους για την παρουσία τους εδώ σήμερα. Με την παρουσία μας, όχι μόνο θα έχουμε ένα συγκροτημένο και διαρθρωμένο διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα και με άλλα θεσμικά όργανα και με την κοινωνία των πολιτών γενικώ. Με την παρουσία μας εδώ σήμερα στέλνουμε και ένα ηχηρό μήνυμα, ένα μήνυμα χειραφέτησης, ένα μήνυμα ε, μη διάκρισης ένα μήνυμα ελευθερίας, όπως μας είπε και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εμείς διεκδικούμε τα δικαιώματά μας. Άνευ όρων ζητούμε να είμαστε πολίτες άνευ όρων. Πολίτες των χωρών μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό το μήνυμα θέλουμε να φτάσει σε όλους τους πολιτικούς ηθήνοντες στα χωριά, στις πόλεις, στις πρωτεύουσες ε, όλων των κρατών μελών και φυσικά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας εύχομαι λοιπόν μια καρποφόρα εκδήλωση και να επισημάνω τίποτα για μας χωρίς τη συμμετοχή μας. Ευχαριστώ. I think I should give Köszönöm szépen. Köszönöm szépen elnök úrnak és az európai ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Κώστας, σας ευχαριστώ πολύ για, το, για την εισαγωγική ομιλία του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Αναπηρίας. Να σας ε, συστηθώ. Είμαι ο Άνταμ Κώσα. Είμαι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είμαι ένας από τους συμπρόεδρους ε, της διακομματικής ομάδας για τα άτομα με αναπηρία. Καλημέρα σα ε, Να σα πω ότι προσεγγίζουμε το 2019, το έτο των ευρωεκλογών, των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι λοιπόν αρκετά επίκαιρη αυτή η συζήτηση της καθολικής ε, χειραφέτησης ε, στα κρατη μελη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς έχει λοιπόν η κατάσταση. Τι γίνεται με το δικαίωμα ψήφου των ατόμων με αναπηρία. Θα το συζητήσουμε το θέμα αυτό λοιπόν σήμερα το πρωί. Και θα κοιτάξουμε μεταξύ άλλων και τα εξή ερωτήματα. Κατά πόσον υπάρχουν ε, φυλάδια τα οποία να είναι προσβάσιμα με άτομα με αναπηρία, να είναι γραμμένα σε ε, σύστημα μπράι, σε φόρμα, σε μορφότυπο το οποίο θα επιτρέπει να το διαβάσουν άτομα με αναπηρία. Έχουν αρρωγή τα άτομα με αναπηρία για να ψηφίσουν και πώς ε, μπορούμε να άρουμε τα εμπόδια για άτομα τα οποία θέλουν να κατέβουν ως υποψήφοι. Πρέπει να αναθεωρήσουμε μήπως ε, τους νόμους για τη νομική για τη δικαιοπραγματική ικανότητα. Καταρχάς λοιπόν οι εμπειρογνώμονες θα έχουν την δυνατότητα να πάρουν το λόγο. Θα έχουν ε, πέντε λεπτά στην διάθεσή τους και θα ήθελα να σας επισημάνω ότι έχουμε χρονική πίεση. Θα ήθελα να τηρείτε όλοι το χρόνο σας. Έχουμε μία ώρα για τους εμπειρογνώμονες και θα ήθελα να βγάλουμε 10 λεπτά από την ώρα αυτή για να ακούσουμε και ερωτοαπαντήσεις. Και μετά την πρώτη εισαγωγή, οι εμπειρογνώμονες θα έχουν από δύο λεπτά στην διάθεσή τους. Έχουμε ένα κατάλογο με τους ομιλητές και θα προεδρεύσουμε με τους συμπροέδρους ε, τις συζητήσεις. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που θέλουν να πάρουν το λόγο και ως εκ τούτου θα σας ζητούσα να τηρείτε το χρόνο ομιλία σας. Θα σας κάνω προφανώς και ε, μήνυμα εάν τελειώνει ο χρόνος σας. Θα ήθελα να συζητήσω στο σημείο αυτό να συζητήσω τον συνάδελφο Μάρκ Πλούρα και την κυρία Πιγκό. από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Αναπηρίας. και θα ήθελα να πάρω και αυτό το λόγο. Ε, κατά εξαίρεση θα ήθελα να δώσω το λόγο ε, συντομία στον πρώτο μας ε, εμπειρογνώμων, τον κύριο Γιώργιο Ντάση, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, ο οποίος πρέπει να μεταβεί δυστυχώ σε μια κηδεία στι 10.30 ενό συναδέλφου. Γι' αυτό λοιπόν θα του δώσω το λόγο κατά εξαίρεση. Δεν τον βλέπω. Πού βρίσκεται. Α, μόλις ενημερώθηκα ότι δυστυχώς ε, ε, αποχώρησε, δεν μπορούσε να παραμείνει δυστυχώς γιατί και εμείς είχαμε καθυστέρηση στο πρόγραμμα. Μάλιστα. Ωραία. Να αλλάξουμε λοιπόν και να περάσουμε στο δεύτερο εμπειρογνώμονα. Θα ήθελα επ' ευκαιρία να δώσω στην, το λόγο στους συναδέλφους. Καταρχάς ο κύριος Μάρεκ Πλούρα να σας καλωσορίσει με λίγα λόγια. Και στη συνέχεια, μετά τον Μάρεκ Πλούρα, το λόγο θα πάρει η κυρία Πιγκό. Για να σας καλωσορίσουμε. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τους εμπειρογνώμονες. Ο κύριος Πλούρα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ αγαπητέ Άνταμ. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας καλωσορίσω θερμότατα σε αυτή την εκδήλωση Ξέρω πόση μεγάλη προσπάθεια χρειάζεται να καταβάλλετε για να έρθετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να μας παρουσιάσετε τις εμπειρίες σας και να λάβετε μέρος στη συζήτηση αυτή. Και ευχαριστώ και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία για την οργάνωση της σημερινής βαρισιμάτης εκδήλωσης. Χαίρομαι ιδιαιτέρως για την ευκαιρία που έχω να συναντηθώ μαζί σας. Χαίρομαι πραγματικά ότι θα συντονίσω και αυτό το πάνελ που για μένα έχει ιδιαίτερη σημασία. Γιατί είμαι άτομο με αναπηρία και όπως όλοι εδώ στην Ομίγυρη είμαι και ψηφοφόρος και μάλιστα ήμουν και υποψήφιος ε, στις ευρωεκλογέ και έχω γίνει και ευρωβουλευτής. Για πολλά χρόνια ενεργοποιήθηκα ε, σε προσπάθειες ε, αποκατάσταση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και εξασφάλιση του δικαιώματος του εκλέγην και του εκλέγεσθε για τα άτομα με αναπηρία. Είχαμε πολλές επιτυχίες ε, στην Πολωνία και καταφέραμε να ε, εξασφαλίσουμε την αναγνώριση, την αναγνωρισιμότητα του φόρου μας και να προωθήσουμε τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Και πραγματικά οι εμπειρίες της πολωνικής αντιπροσωπής ήταν πολύ θετικές. Δυστυχώς ε, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια ανησυχητική πορεία στην Πολωνία, μια προσπάθεια επαναχώρηση σε σχέση με τα πολύ σημαντικά αυτά δημοκρατικά επιτέγματα. Γι' αυτό και θέλουμε να αναχαιτήσουμε αυτή την προσπάθεια παλιδρόμησης σε σχέση με τα δικαιώματα. Όχι, θα πρέπει να διεκδικήσουμε, να συνεχίσουμε να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας. Και πιστεύω ότι σε πολλά κράτη-μέλη έγιναν αλλαγές ε, επιτρέποντας σε εκατομμύρια συμπολίτες μας ε, με αναπηρία να απολαύσουν τα δικαιώματά τους, τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητα του πολίτη. Και χαίρομαι που σήμερα θα ακούσουμε τις βέλτιστες πρακτικές στην συζήτηση αυτή. Βέβαια, είμαι πεπισμένος ότι πολλά ακόμη θα πρέπει να γίνουν. Πάντως, η Ευρώπη χρειάζεται και τη δική μας φωνή, χρειάζεται και τη δική μας ψήφο, χρειάζεται και τη δική μας συμμετοχή στον πολιτικό βίο, στις συζητήσεις, στη διαμόρφωση των πολιτικών προγραμμάτων και πάνω απ' όλα στη λήψη αποφάσεων. Και γι' αυτό η σημερινή εκδήλωση θα μας βοηθήσει να εντοπίσουμε τους φραγμούς στα εμπόδια και να προτείνουμε λύσεις, ώστε η αναπηρία να μην περιορίζει τα δικαιώματα του πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά εν είδη εισαγωγής. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην συμπρόεδρο επίσης αυτού του τμήματος της συζήτησης, στην κυρία Μωρίν Πιγκό, που είναι μέλος εκτελεστικής επιστροπής του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπήρεια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πλούρα, και είναι μεγάλη μου μεγάλη μου τιμή που συμμετέχω στι σημερινές συνεδριάσει και στη σημερινή εκδήλωση. Προσφάτως εκλέχθηκα στην Εκτελεστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για άτομα με αναπηρία και σε ό,τι αφορά και την Ένωση των ατόμων με διανοητική αναπηρία και τι οικογένειε τους. Σήμερα είναι ιστορική ημέρα όπως μας ε, είπε και ο συνάδελφος, κλείνουμε 10 χρόνια από την υπογραφή της συνθήκης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία από τους ηγέτες όλου του κόσμου σε επίπεδο ΟΗΕ και 20 χρόνια από τότε που ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία για να έχουμε έναν τρόπο να συνεργαζόμαστε, να ενώσουμε τις φωνές μας για όλα τα άτομα με αναπηρία σε όλη την Ευρώπη. Είναι επίσης ιστορική ημέρα γιατί έχουμε την ευκαιρία να καταστήσουμε την επόμενη δεκαετία μια εντελώς διαφορετική δεκαετία. Και θεωρώ επίσης ότι είναι ιστορική η σημερινή ημερομηνία λόγω της τεράστιας προσέλευσης που έχουμε εδώ. Περίπου 800 άτομα με αναπηρία από όλα τα, όλες τις γωνιές της Ευρώπης που εκπροσωπούν την πλήρη ποικιλομορφία των ατόμων με αναπηρία στην Ευρώπη και είμαι απόλυτα ενθουσιασμένοι και έκθαμβοι που από αυτούς τους 800 περίπου 200 είναι άτομα με διανοητική αναπηρία γιατί πραγματικά αυτό είναι κάτι το καινούργιο, το προποριακό, το ιστορικό. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό ότι υπάρχει όλο και με πιο μεγάλη αποφασιστικότητα από τα άτομα με αναπηρία να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Αυτό είναι κάτι το ενθαρρυντικό. Κάτι το ενθαρρυντικό για τα άτομα αυτά τα οποία ακόμα και τα άτομα αυτά τα οποία ιστορικά ήταν τα πιο απομονωμένα και αυτό σημαίνει ότι έχουμε τρόπους να συνεργαστούμε και να βρούμε εταίρους και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες μας γιατί όλα αυτά λειτουργούν γιατί όλοι έχουν έρθει μέσω των εθνικών αντιπροσωπιών τους με υποστήριξη των Ευρωβουλευτών και εξ ονόματος των οργανώσεων και των ενώσεων που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία. Έχουμε βρει λοιπόν τρόπους να συνεργαζόμαστε, να δημιουργούμε συμμαχίες, εταιρικέ σχέσεις. Αυτή είναι η πολιτική ενδράση. Αυτή είναι η πλήρη συμμετοχή στις ευρωπαϊκές, στο ευρωπαϊκό πολιτικό γίγνεσθε. Αλλά έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε υπάρχουν ακόμα άτομα τα οποία δεν μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Με μια τέτοια σκληρή απόρριψη υπονομικής άποψης ως ανθρώπινα όντα. Τους αρνούνται την δικαιοπρακτική τους ικανότητα, την ε, πλήρη ευθύνη για τον εαυτό τους και αυτό στερεί από κάποιους ανθρώπους το δικαίωμα τους να δρουν εξ ονόματός τους, να τους παίρνουν στα σοβαρά όλα τα θεσμικά όργανα της κοινωνίας. Και αυτό είναι επονίδιστο το 2017 στην Ευρώπη να υπάρχει μια τέτοια κατάσταση. Μέχρι ότου μεταρρυθμίσουμε λοιπόν τους νόμους αυτούς, μέχρι ότου καθιερωθεί το δικαίωμα για τη λήψη αποφάσεων και μέχρι και το σημείο που και ο τελευταίος άνθρωπος δεν θα είναι ελεύθερος στην κοινωνία μας, δεν θα είναι κανείς ελεύθερος. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε ως κίνημα. Επίσης, ακούσαμε και για τα άλλα εμπόδια τα οποία θα πρέπει να αφαιρεθούν. Αν σημειωθεί επιτυχία λοιπόν σήμερα, θα πρέπει να σημειωθεί μία διαφορά. Και μέχρι το επόμενο φόρουμ για τα άτομα με αναπηρία στο Κοινοβούλιο θα διαπιστώσουμε ότι πρόκειται για την αρχή της νέας αυτής δεκαετίας που περιγράφησε ο Γιάννη. Και τι διαπιστώνουμε ότι η, ε, θα διαπιστώσουμε ότι οι ευρωεκλογέ το 2019 θα είναι προσβάσιμες και ότι θα συμμετέχει ο κόσμος σε μεγάλο ποσοστό και ότι θα εκλεχθούν πολλά τέτοια άτομα εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο και θα έλθουν να συνεργαστούμε τους συναδέλφους τους. Τι άλλο θέλουμε να δούμε. Θέλουμε να δούμε και ένα ευρωπαϊκό έτος ατόμων με αναπηρία, ένα πολυετές ε, πρόγραμμα και προϋπολογισμός ε, προκειμένου να υπάρχει συμπερίληψη σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα πρέπει να δούμε ότι όταν θα γίνει η επόμενη μελέτη από τη ΦΡΑ για το 2022 θα προκύψει ότι δεν θα υπάρχει καμία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου ο κόσμος δεν θα έχει δεν μπορεί να ασκεί τα βασικά αυτά τα δικαιώματα. Είναι λοιπόν καθήκον μας σήμερα να συνεργαστούμε με τους ευρωβουλευτές που μας κάλεσαν σε, σε αυτή την ιδιαίτερη εκδήλωση που μας εμπνέει να συνεργαστούμε με τους επιτρόπους και να βρούμε τρόπους συνεργασίας με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και στη συνέχεια να επανέλθουμε στις πόλεις μας, στις κοινότητές μας, στις χώρες μας ο καθένας και να απαιτήσουμε να συμπεριληφθούμε, να δώσουμε εκπαίδευση, κατάρτιση στον κόσμο για το πώς μπορεί να ασκεί πλήρως τα δικαιώματά τους ως πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης χθε συναντηθήκαμε με την Ένωση για την ε, αυτό εκπροσώπηση στην Ευρώπη και το μήνυμά τους ήταν ξεκάθαρο και σαφέστατο. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ενωμένοι στα σαφή και ξεκάθαρα δικαιώματα που απαιτούμε για τα άτομα με αναπηρία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Πιγκό για την εισαγωγική σας αυτή ομιλία. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο ε, στον πρώτο μας εμπειρογνώμονα, τον Χάρη Ρος, και να τον παρακαλέσω να τηρήσει το πεντάλεπτο που είναι ο χρόνος αγόρευσης για τους εμπειρογνώμονές μας και τους καλεσμένους. Good morning. Καλημέρα σας. Αγαπητοί προβουλευτέ, ε, μέλη της Επιτροπής, λένε στον ομιλητή να μην πλησιάζω πολύ στο μικρόφωνο γιατί μπουκώνει. Ξαναρχίζω. Καλημέρα σας, Ευρωβουλευτές, μέλη της Επιτροπής, ε, υπάλληλοι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής και ε, μέλη των ε, φορέων που εκπροσωπούνται σήμερα εδώ είναι μεγάλη μας τιμή να βρισκόμαστε εδώ. Ονομάζομαι Χάρη Ρόουτς και είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Inclusion Europe δηλαδή ε, ένταξε στην, και ενσωμάτωσε στην Ευρώπη για δικές ανάγκες είναι ε, σε μια πλατφόρμα του Ηνωμένου Βασιλείου και ασχολούμαι εκεί στο Διευθυντικό Συμβούλιο, τόσο ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε κάποιους που έχουν ε, διανοητικά προβλήματα να μπορέσουν να έχουν το δικαίωμα του και του εκλέγεστε. Επίσης θα πρέπει να δούμε τι προβλέπει η σύμβαση του ΟΗΕ για τα πρόσφατα αναπηρία, τι θα πρέπει να κάνουν οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό επίσης έχω προσωπικά παραδείγματα, προσωπικές εμπειρίες για το ότι μπορεί κάποιος να συμμετάσχει στον πολιτικό γίγνεσθε στην πατρίδα μας, αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα. Τέταρτον, να δούμε το πώς ε, όλοι όσοι παριστάμεθα σήμερα εδώ μπορούμε να κάνουμε την ε, διαφορά. Είτε εργαζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είτε ε, εργαζόμαστε στα πλαίσια μιας οργάνωσης προσώπων με αναπηρία. Τι αποτελεί φραγμό στο δικαίωμα του εκλέγει αυτά τα πρόσωπα. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται ε, όσον αφορά τον αστικό κώδικα των χωρών για τη δικαιοπρακτική ικανότητα αυτών των προσώπων γιατί πολλές φορές ζουν σε κάποια ιδρύματα ε, αυτά τα πρόσωπα και δεν μπορούν να ψηφίσουν. Και σε πολλές χώρες δεν μπορούμε να έχουμε το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε, δεν μπορούμε δηλαδή και μέλη κάποιων φορέων, δεν μπορούμε να λάβουμε κάποιο αξίωμα. Και εξηγώ με ένα παράδειγμα, μία γυναίκα στην Ισπανία θα έπρεπε να περάσει κάποιες ε, εξετάσεις για να αποδείξει ότι μπορεί να ψηφίσει. Και επίσης σας ε, ρωτώ, μα τι θα γινόταν εάν όλοι θα πρέπει να περάσουν εξετάσεις για να ψηφίσουν, πόσοι ψηφοφόροι θα περνούσαν αυτές τις εξετάσεις και με μεγάλη μου χαρά διαπιστώνω ότι όλα τα κόμματα που προσωπούνται στην Ισπανική Βουλή υποσχέθηκαν ότι αυτός ο νόμος θα καταργηθεί. Ακόμη και αν ε, το δίκαιο, αν ο νόμος δεν μας απαγορεύει το να ε, ψηφίσουμε, η προσβασιμότητα παραμένει μεγάλο πρόβλημα στα εκλογικά τμήματα. Ε, έχουν γίνει τέτοιες ρυθμίσεις που μας ε, δυσκολεύουν ή δεν μπορούμε να καταλάβουμε το πώς λειτουργεί αυτή ρύθμιση. Θα πρέπει να δούμε το πώς θα γραφούμε στους εκλογικούς καταλόγους, το, ποιον και πώς θα ψηφίσουμε. Όλα αυτά είναι αρκετά δύσκολα, περίπλοκα και δεν υπάρχουν κάποιου είδου κατανοητές, της οδηγίες και οι, όσοι εργάζονται στα εκλογικά κέντρα δεν βοηθούν τους ε, αναπήρους ε, ψηφοφόρους και πάρα πολλές φορές τα πρόσωπα που έχουν διανοητικά προβλήματα δεν προσκαλούνται ε, σε συναντήσει πολιτικού χαρακτήρα, σε πολιτικέ συγκεντρώσει. Δεν του ρωτάει κανεί τη γνώμη του για τα βασικά προβλήματα στην κοινότητα όπου ζουν. Υπάρχουν επίση κάποιε προκαταλήξει για αυτέ τι διανοητικέ δυσκολίε ε, και έτσι είναι πιο δύσκολο αυτά τα πρόσωπα να συμμετάσχουν, να μπορούν να αποκτήσουν κάποια εμπειρία και να προβάλλουν τι δεξιότητέ του τι ικανότητέ του και αυτό ε, αφορά και τα μέλη τη οικογένεια του πολλοί που ζουν σε κάποια ιδρύματα που είναι πλαισιωμένοι κάποιες φροντίδες δεν μπορούν να γραφούν στο κληρικό κατάλογο ή να ψηφίσουν. Ακόμη και το να πάνε στο κληρικό τμήμα αποβαίνει δύσκολο. Ο οφόρια μας, CRPD, είναι μια επιτροπή και ε, θέλουμε να δούμε τι γίνεται με αυτή την εφαρμογή της συνθήκης του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης να δούμε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση τα πρόσωπα με αναπηρία ε, θα πρέπει να έχουν πλήρη δικοπατικά ικανότητα, δικοπατικά ικανότητα ιδίως εκείνοι που ζουν στο ίδρυμα να μπορούν να έχουν πρόσβαση δηλαδή στο χώρο της ψηφοφορία και επίσης η Επιτροπή μας, ο φορέας η, η, η σύμβαση CRPD λέει ότι όλοι που έχουν να πειρήσετε πρέπει να έχουν αυτά όλα τα δικαιώματα ακόμα και αυτοί που τελούν υπό κάποιο είδου ε, κυδαιμονία, επιτροπία ε, και επίση να μπορεί να υπάρχει επικοινωνία, να υπάρχουν σχετικές διευκολύνσεις. Τι μπορεί να γίνει για να βελτιωθεί αυτή η προσβασιμότητα. Η ManCap, ο φορέας μας, κάνει μια εκστρατεία, διακόπτη πρόεδρος. Κοιτάξτε, επειδή πιεζόμαστε από τον χρόνο θα πρέπει να συντομεύσετε κάπως. Καλώς, καλώς Μωρίνη, σε ευχαριστώ λέει ο κύριος Ρόουτς προς την πρόεδρο. Ναι, πρόκειται και το θέλουμε να μπορούν ε, οι άνθρωποι με αναπηρίες να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους και πάρα πολλοί πολιτικοί δεν ξέρουν ποια είναι τα προβλήματα των ανθρώπων που έχουν διανοητικές δυσκολίες. Επίσης, θα σας παραθέσω κάποια παραδείγματα κάποιων συγκεκριμένων πολιτικών οι οποίοι είχαν ε, διανοητικά προβλήματα η Σάρα Πίκαλ έχει εκλεγεί στην κοινότητά της επί έξι ε, χρόνια ως ε, μέλος της αυτοδιοίκησης και είναι περήφανη που προσωπεί ε, όσους ε, έχουν προβλήματα τέτοια και όμως προσωπούνται τώρα στο αυτό συμβουλίο. Επίσης στην Ισπανία γίνεται το ίδιο και η Άγχελα μπήκε στην πολιτική τον ε, Μάιο του 2011. Το 2015 ο Γκάβιν Χάρντινγκ έγινε δήμαρχος του Σέλμπι στο βόρειο Yorkshire. Το 2014 βραβεύτηκε από τη Βασίλισσα για τις υπηρεσίες του υπέρ των ε, ανθρώπων με αναπηρία. Να, προγράμματα κάποιων που έχουν αναπηρίες και ξεπέρασαν τους σχετικούς φραγμούς. Εξελέγησαν και συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων. Χάρη σε ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Thank you, Harry. I'm sorry, I know you were told you had very hard to cut a presentation. Thank you. Σε ευχαριστώ θερμά γιατί ξέρω πόσο δύσκολο είναι να πρέπει να, να συντομεύσει κανείς την ομιλία που έχει προετοιμάσει. Ο κύριος Πλούρα, σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ χρήσιμη και πολύ σημαντική για όλους σας η ομιλία μας. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Δημήτρη Παπαδημούλη, Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και μάλιστα είναι και πρόεδρος της ομάδας υψηλού επίπεδου για την ισότητα των δύο φύλων και επίσης έχει, α, έχει, δεσμευθεί υπέρ του ανοίγματο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να γίνει πραγματικά ανοιχτό θεσμικό όργανο. Συγγνώμη, ε, κύριε Παπαδημούλη. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη α, γιατί το σύστημά μας δεν λειτουργεί πάντα εύκολα. Αυτό το σύστημα με τους υποτίτλους έχει μια υστέρηση χρονική. Θα προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε Βαρδακαστάνη, κύριοι ε, συμπρόεδροι, μέλη της διακομματικής ομάδας για τα άτομα με αναπηρία, ε, κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές, μέλη της διοίκησης, ε, αγαπητοί φίλοι Νιώθω μεγάλη χαρά που συμμετέχω σήμερα στο τέταρτο Ευρωκοινοβούλιο των ατόμων με αναπηρία. Με βάση τα στοιχεία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα στου έξι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάποια αναπηρία, ήπια σε ω σοβαρή μορφή. Περίπου 80 εκατομμύρια συμπολίτε μα είναι συνολικά τα άτομα με αναπηρία. Πριν από λίγε μέρε, πριν από τρει μέρε. η 3η Δεκεμβρίου ήταν η Διεθνής διεθνή μερα των Ατόμων με Αναπηρία. Ε, εορτάζουμε αυτή τη μέρα για να προωθήσουμε ε, την στήριξη των ατόμων με αναπηρία και να ε, συνειδητοποιήσουμε όλοι τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν αυτά τα άτομα. Και μάλιστα χαίρομαι που εορτάζουμε αυτή τη μέρα με την ε, ε, οργάνωση μιας ενημερωτικής συνεδρίασης για τα μέλη του προσωπικού και τα άτομα που έχουν στην οικογένειά τους κάποιον άνθρωπο με αναπηρία. Επίσης, έχουμε την ομάδα υψηλού επίπεδου ε, ισότητας και πολυμορφίας ε, τις οποίες προεδρεύω και έχουμε δεσμευτεί υπέρ της πλήρους εσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρία. Θέλουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γίνει ένας χώρος που θα είναι απόλυτα προσβάσιμος σε όλους. Ήδη το 2006 το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υιοθέτησε μια δήλωση επί της αρχής προκειμένου να προωθήσουμε την ισότητα και την ε, πολυμορφία, τη διαφορετικότητα στη γραμματεία. Αυτός είναι πρωταρχικός στόχος για να ενσωματώσουμε καλύτερα και στο, στην απασχόληση τα άτομα με αναπηρία. Επίση, έχουμε υιοθετήσει το δεύτερο πολιτέ πρόγραμμα δράση για την ισότητα των φύλων και τη διαφορετικότητα που καλύπτει την περίοδο 2014-2019. Αυτό το σχέδιο δράση αποτελεί το βασικό εργαλείο για την υλοποίηση απτή ε, προόδου σε ό,τι αφορά την ισότητα και τη διαφορετικότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και σε ό,τι αφορά τα άτομα με αναπηρίες, ε, το σχέδιο δράσης προβλέπει τέσσερις ε, θεμελιώδεις στόχους. Καταρχήν να αναπτύξουμε την κουλτούρα του θεσμικού οργάνου απέναντι στην αναπηρία, να υιοθετήσουμε κάποια θετικά μέτρα να προωθήσουμε την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία, να διευκολύνουμε την ε, ένταξη στον χώρο εργασία και τη σταδιοδρομία των ατόμων ε, με αναπηρία και να προωθήσουμε την προσβασιμότητα των κτηρίων, των χώρων εργασία και την καλύτερη ενημέρωση των ατόμων με αναπηρία. Επίση, θα ήθελα να τονίσω ότι μέχρι στιγμή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μοναδικό θεσμικό όργανο τη Ευρωπαϊκή Ένωση που ε, προσφέρει θετικά προγράμματα δράση για του υπαλλήλου με αναπηρία. Και μάλιστα τελευταία οι 11 υπάλληλοι έχουν προσληφθεί με κάποια αναπηρία, ε, αποδεικνύοντα και εμπράκτο την προσήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο στόχο αυτό. Επίσης, δίνουμε προτεραιότητα σε θέματα όπω ε, ο συνδυασμό τη ε, προσωπική και επαγγελματική ζωή, η αξιοπρέπεια στον χώρο εργασία και ο σεβασμό του ανθρώπου, όπω φαίνεται από την πολιτική μα για την πάταξη τη παρενόχληση. Μόνο χάρη σε στην ε, συνεργασία όλων και την προσήλωση όλων θα εξασφαλίσουμε συμμετοχή και ενσωμάτωση των ατόμων και αναπηρία παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα συνεχίσω τις προσπάθειές μας ε, προκειμένου να ενθαρρύνουμε και να εξασφαλίσουμε συντονισμό για τη συμμετοχή ε, και την ενσωμάτωση υπαλλήλων με αναπηρία. Σας ευχαριστώ. Bardzo σας ευχαριστούμε κύριε Παπαδημόλη. Όντως έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια μέχρι στιγμής. Πολύ σημαντικό έργο έχει δηλοποιηθεί και πραγματικά έχουμε αποδείξει εμπράκτος ότι το θεσμικό όργανο που εκπροσωπούμε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βρίσκεται στην πρωτοκαθεδρία τέτοιων δράσεων. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον Ξύστο Πάτερ, που είναι μέρος ε, της ΕΟΚΙ, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ε, και εισηγητής ε, της έκθεσης που αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα ε, τα άτομα με αναπηρία. Παρακαλώ, κύριε Ξίστοφ Πάτερ, έχετε το λόγο. Ε, Κυρίες και κύριοι, δεν σκόπευα προφανώ να αφαιρέσω το 50% τη ομιλία μου, αλλά ελπίζω να κατάφερα. Είναι σαφέ ότι για πολλά άτομα με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δικαίωμα ψήφου δεν ε, είναι πραγματικό, αλλά καθαρά θεωρητικό. Εγώ προετοιμάζω την έκθεση τη Ευρωπαϊκή Κοινωνική και Οικονομική Επιτροπή για τα πραγματικά δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία σε ό,τι αφορά την ψήφο του ε, για τι ευρωεκλογέ. Και σκοπό μα είναι να παρουσιάσουμε σε λίγου μήνε μια συνεκτική λεπτομερή ανάλυση για το πώ διαμορφώνεται πραγματικά η κατάσταση, η πραγματικότητα. Αν κάποιο θα ήθελε να μα βοηθήσει συλλέγοντα δεδομένα από οργανώσει και από θεσμικά όργανα στι χώρε του, σα παρακαλώ ε, συμπληρώστε την, ε, το δελτίο, το κίτρινο και πράσινο, το οποίο θα βρείτε έξω και προσθέστε το σας παρακαλώ επικεντρωνόμαστε στις ευρωεκλογέ, αλλά είμαστε βέβαιοι ότι η πρωτοβουλία για τη βελτίωση των, της νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα επηρεάσει και την νομοθεσία σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για τις εθνικές και περιφερειακές εκλογές. Πιστεύω ότι η, όταν θα περάσει η έκθεση αυτή, οι πολιτικοί θα έχουν ε, στη διάθεση τις πληροφορίες που χρειάζονται για να πάρουν αποτελεσματικά μέτρα. Δεν θα υπάρχει πλέον περιθώριο για δικαιολογίε. Όντως, οποιαδήποτε αλλαγή για το εκλογικό δίκαιο στο ευρωπαϊκό επίπεδο προαπαιτεί ομόφωνη απόφαση των κρατών μελών, αλλά επίση αληθεύει ότι δεν πρέπει να συμβεί τίποτα έω ότι περάσουν αυτέ οι προτάσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και άρα, αγαπητό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι η δική σα σειρά να κάνετε το επόμενο βήμα, χωρί να περιμένουμε την τελευταία έκθεση, την τελευταία ε, μορφή τη έκθεση. Ξέρουμε ήδη ότι σε κάθε κρατό μέλος θα πρέπει να σημειωθούν βελτιώσει στην νομοθεσία και πολλές χώρες όπως σας αναφέρθηκε ουσιαστικά αφαιρούν κάποιες ομάδες αυτόματα από τη συμμετοχή στις πολιτικές ομάδες και το δικαίωμα ψήφου για πολύ κόσμο είναι αφαιρείται σε πολλέ περιπτώσεις. Αυτό ισχύει σε 11 κράτη-μέλη. Σε 7 άλλα κράτη-μέλη το δικαστήριο έχει δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση στην ψηφοφορία, στη συμμετοχή σε ψήφο, ε, σε περίπτωση που αποφανθεί έτσι. Και σε άλλα κρατημέλη μπορεί λόγω αναπηρίας να αρνηθεί κάποιος ένα άτομο με αναπηρία να ψηφίσει. Αλλά ακόμα και σε χώρες που δεν έχουν τέτοιους περιορισμούς υπάρχουν εκατοντάδες εμπόδια που εμποδίζουν σε εκατομμύρια ανθρώπους να ψηφίσουν. Να πω μερικά από αυτά στην σύντομη παρουσίασή μου σε πολλά κράτη-μέλη κανείς δεν φροντίζει το φόρουμ για την ε, παροχή πληροφοριών, τη μορφή των ε, παροχής πληροφοριών στα άτομα αυτά. Και αυτό αποτελεί μεγάλη πρόκληση και επίσης το πώς μπορεί να μεταβεί κανείς στα εκλογικά κέντρα ε, προβλήματα πρόσβασης για τα άτομα με αναπηρία, με κινητική αναπηρία. Άλλο πρόβλημα μέσα στα εκλογικά κέντρα πλέον, σε πολλά εθνικά συστήματα υπάρχουν νομικές διατάξεις που περιορίζουν σημαντικά την αρρωγή που παρέχεται από προσωπικούς βοηθούς ή που υποχρεώνουν τους ε, ψηφοφόρους να ζητούν βοήθεια από τους ε, υπαλλήλου στο εκλογικό δικαίωμα. αντίθετα με την εμπιστευτικότητα και επίσης ε, τίθεται το θέμα του τόπου κατοικία. Αυτό σε πολλέ περιπτώσει σημαίνει ότι δεν έχει ο κόσμο δυνατότητα να ψηφίσει. Επίση, πολλά προβλήματα σε ό,τι αφορά τα δελτία. Αυτά τα αναφέρω στην εκθεσή μου επισταμένω. Καταλαβαίνω ότι θα πάρει χρόνο να εγκαθιδρυθούν τα πραγματικά πλήρη δικαιώματα ψήφου για όλα τα άτομα με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά τώρα πρέπει να πούμε ότι οι διατάξει που εμποδίζουν τα άτομα με αναπηρία να ψηφίσουν λόγω σωματική ή δυνητικής αναπηρία θα πρέπει να καταργηθούν άμεσα. Όλοι οι πολίτε συμπεριλαμβανομένων αυτών που δεν μπορούν να μεταβούν καν στο εκλογικό κέντρο, θα πρέπει να έχουν δικαίωμα, πραγματικό δικαίωμα ψήφου. Και οι σχετικέ διατάξει θα πρέπει να επιτρέπουν σε όλα τα άτομα να ψηφίζουν αυτοπροσώπως και με εμπιστευτικότητα, με απόρριτο. Αυτό αφορά, ξέρετε, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε διατάξει που δεν εγγυώνται αυτό το δικαίωμα για εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες. Έχει έρθει η στιγμή να το αλλάξουμε και έχουμε ακόμα χρόνο πριν από τις ευρωεκλογέ το 2019. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε κύριε Ξίστοφ Πάτερ. Πραγματικά πολύ σημαντική έκθεση που εκπώνησες και που δίνει κάποιες συστάσεις ε, για τις μελλοντικές δράσεις που απαιτούνται. Ε, και ε, θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Πίγκοτ, την εκτελεστική διευθύντρια, για να δώσει το λόγο στον επόμενο ομιλητή, τον Πατ Κλάρκ, που είναι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία. Παρακαλώ, κύριε Κλάρκ, έχετε το λόγο. Καλημέρα σε όλους. Ο κύριος Κλάρκ. Ευχαριστούμε που μας προσκαλέσατε. Είναι πολύ σημαντική υπόθεση που σήμερα μας απασχολεί και ελπίζουμε να, να αυτό που θα πούμε είναι στο ύψος των περιστάσεων. Έχουμε το μανιφέστο του EDF όσον αφορά τις ευρωεκλογές του 2019. Εισαγωγικά να σας πω ότι φέτος το EDF συμπληρώνει 20 χρόνια ύπαρξης και έχουμε εσάς τους εκπροσώπους των ανθρώπων με αναπηρίες από το αναπηρικό κίνημα. Και όταν συντάξαμε αυτό το μανιφέστο για τις ευρωεκλογέ, είχαμε κατά νου τα εξή. Θέλουμε να υπάρχουν ευρωεκλογέ οι οποίε να ενσωματώνουν τους πάντε και καλούμε τους Ευρωπαίους ηγέτε να φροντίσουν ούτω ώστε οι άνθρωποι με αναπηρία να συμμετέχουν στι εκλογέ και να γίνουν τα εξή. Θα πρέπει οι άνθρωποι με αναπηρίε να έχουν δικαίωμα εκλέγει και εκλέγεστε ακριβώς όπως προβλέπει το άρθρο 29 της Σύμβασης CRTD. Θέλουμε να τροποποιηθεί η νομοθεσία για τη διοικητική ικανότητα σύμφωνα με τη συνθήκη θέλουμε στα εκλογικά τμήματα, εκλογικά κέντρα να μπορούν όλοι να πάνε και επίσης τα των εκλογών να είναι πιο εύχοστα, πιο κατανοητά και να υπάρχουν όλες οι διευκολύνσεις να μπορούν να συμμετάσχουν ε, οι άνθρωποι με αναπηρίες σε συζητήσεις, σε ιστοσελίδες και επίσης ε, να ε, υπάρξει σωστή δεδομένων για την πολιτική συμμετοχή και ανάλυση να δεδομένων αυτόν για τα πρόσωπα με αναπηρία. Και επίσης θέλουμε να υπάρχει μια στρατηγική, σφαιρική, συλλογική και χαιρετίζουμε την δέσμευση για τις υποσχέσεις του Πρόεδρου Ταγιάννη να υπάρξει μια στρατηγική 2020-2030 για τους ανθρώπους με αναπηρία σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση και επίσης να υπάρξει και προϋκοδότηση για την εφαρμογή της. Να υπάρξει συνέχεια στη στρατηγική 2020 επί τη βάση των συμπερασμάτων που έχουν εξαχθεί από την ε, Επιτροπή του ΟΗΕ για την Ευρωπαϊκή Ένωση στους ανθρώπους με αναπηρία και αυτό να ληφθεί υπόψη από κάθε θεσμικό όργανο και με μια τέτοια στρατηγική να μπορέσουμε να προωθήσουμε την ιδέα ενός θεματολογίου και το 2021 να είναι η χρονιά των ανθρώπων με αναπηρία και επίσης τότε να εορταστεί η συμπλήρωση δεκατών από την σύμβαση του ΟΗΕ να μην υπάρχουν δυσμενείς διακρίσεις να υπάρχουν ε, κάποιες εξασφαλίσεις για μια συνεκτική πολιτική που να ενσωματωθεί στην, στην πολιτική που θα ασκείται και να χρησιμοποιήσουμε και να αξιοποιήσουμε τα διαφορετικά ταμεία ούτω ώστε να μπορέσουν ουσιαστικά να συμμετάσχουν οι οργανώσεις ε, των ανθρώπων με αναπηρία στην διαμόρφωση του προϋπολογισμού επίσης και στους κοινωνικούς πυλώνες να ε, ε, υπάρξουν κατάλληλες ε, ρυθμίσεις και να υλοποιηθούν αυτές. Θέλουμε εφαρμογή του κοινωνικού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και των σχετικών πρωτοβουλειών. Να υπάρξει μια πλατφόρμα για τις οικογένειες των ανθρώπων με αναπηρία, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί αξιοπρεπής διαβίωσή τους να εξασφαλιστεί επίσης η απασχόληση των προσώπων αυτών, να υπάρξουν προγράμματα και νομοθεσία όσον αφορά την απασχόλησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι όσοι έχουν αναπηρία να έχουν το δικαίωμα σε μια ε, παιδεία που τους εντάσσει σε αυτήν. Να μην ε, απομονώνται σε ιδρύματα. Θέλουμε οι πολιτικοί οι ηγέτες να εφαρμόσουν την νομοθετική πράξη για την προσβασιμότητα των ανθρώπων με αναπηρία, συνεργασία επίσης για την ε, εφαρμογή της Συμφωνίας του Μαρακές τα βιβλία να έχουν ομορφότυπους που να τα κάνουν προσβάσιμα στους ανθρώπους με αναπηρία και να έχουμε κάποιες πολιτικές ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι τεχνολογικές πρόοδοι δεν θα μένουν μακριά από κανένα να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να απολαμβάνουν την πρόοδο όπως όλοι οι άλλοι. Να μπορούν να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν σε κάθε πτυχή της ε, ζωής. Δικαιώματά τους επίσης να εξασφαλιστούν ως επιβατών. Να μπορούν να έχουν ελευθερία κίνησης και διακίνησης όπως όλος ο κόσμος. Θέλουμε μια Ευρώπη ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει οι πολιτικοί ηγέτες να θεσπίσουν κάποια οριζόντια νομοθεσία για την ισότητα. Να ληφθούν υπόψη επίσης και τα δικαιώματα των ε, γυναικών κάθε ηλικία. Το δικαίωμα στην ισότητα. Να καταπολεμηθεί η βία όπως προβλέπει η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης να σταματήσει η αναγκαστική στήρωση των γυναικών αυτών και σας προτείνω αυτό το κείμενο για έγκριση. Thank you, Pat. ευχαριστούμε, Πατ. Θα έχουμε όλη την ευκαιρία να εγκρίνουμε το μανιφέστο αφού ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Πύρκο Μαλεμάκη από το Φιλανδικό Φόρουμ για τα άτομα με αναπηρία για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Εκ μέρους του Φιλανδικού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία θα ήθελα να απευθύνω ένα μήνυμα στους πολιτικούς ευθύνων της Ευρώπης και στο ευρωπαϊκό αναπηρικό κίνημα. Θα πρέπει να συνεργαστούμε και να μεριμνήσουμε ώστε τα άτομα με αναπηρία να έχουν πλήρες δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεστε στις ευρωεκλογέ. Οι επόμενες ευρωεκλογέ θα είναι οι πρώτες εκλογές μετά την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Θα έχουμε μια ιστορική ευκαιρία να εξασφαλίσουμε πλήρη συμμετοχή και πλήρη εσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία στις ε, ευρωεκλογές ισότιμα με όλους τους υπόλοιπους πολίτες με βάση του άρθρου 29 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές ε, στις εθνικές νομοθεσίες που θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με το άρθρο 12 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των ΑΜΕΑ και επίσης με το Γενικό Σχόλιο 1 της Επιτροπής των ε, ε, Ηνωμένων Εθνών. Δηλαδή θα πρέπει να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ στα εκλογικά κέντρα. Επίσης, ε, η διαδικασία της ψηφοφορίας θα πρέπει να είναι προσβάσιμη για τα άτομα με αναπηρία και θα πρέπει οι ψηφοφόροι να μπορούν να κατανοούν αυτή τη διαδικασία. Έτσι χρειάζονται κάποιες ε, ενημερωτικές εκστρατείες, ε, πολιτικές ε, συναντήσεις, η προσβασιμότητα των ιστοσελίδων και φυσικά και τα έντυπα ή τα άλλα φυλάδια και ψηφοδέλτια να είναι κατανοητά θα πρέπει να μπορούν να ασκούν ανεξάρτητα το δικαίωμα του εκλέγην τα άτομα με αναπηρία. Σήμερα εορτάζουμε την εκατοστή επέτειο της ανεξαρτησίας μας. Πριν από 111 χρόνια οι γυναίκες της Φιλανδίας απέκτησαν δικαίωμα ψήφου και είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε και το δικαίωμα του εκλέγης στους νέους μας. Θα πρέπει και αυτοί να συμμετέχουν στις εκλογές. Ευχαριστώ. Thank you very much. Η κυρία Πίγκοτ, ευχαριστούμε Πίρκο. Στόρκετ Όλισον τώρα από την Δανική Αναπηρική Οργάνωση. Is it on now? Yes. Thank you very much. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω Ευχαριστούμε για την οργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Ξέρω πόσο δύσκολη είναι, ε, πόσο δύσκολο είναι οργανωτικά αυτό το εγχείρημα και πόσο κοστίζει μερικές φορές ακόμη και η έλευση εδώ των ε, συναδέλφων, των συμμετεχόντων. Στη Δανία η κατάσταση για τα άτομα με αναπηρία έχει βελτιωθεί αισθητά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι ιδεώδης θα πρέπει να εξασφαλίζεται η πρόσβαση στις πληροφορίες ε, των πολιτικών κομμάτων. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η συμμετοχή μας στις ε, δημόσιες συζητήσεις. Πολλές φορές γίνονται πολιτικές αναμετρήσεις ε, στην τηλεόραση χωρίς διερμηνία στην νοηματική ή χωρίς υποτίτλους. Πώς είναι δυνατόν ένα άτομο με αναπηρία να παρακολουθήσει τέτοιες τηλεοπτικές πολιτικές αναμετρήσεις. Για να καταφέρουμε όμως να ψηφίσουμε με πλήρη γνώση της κατάστασης θα πρέπει και η ενημέρωσή μας να είναι κατάλληλη. Σε πολλές περιπτώσεις, σε πολλές κοινότητες παρεμποδίζονται τα άτομα με αναπηρία από την υποβολή της υποψηφιότητάς τους στις εκλογές. Είναι απαράδεκτο να μην μπορούμε να σκίσουμε το δικαίωμα του εκλέγεσθε λόγω της αναπηρίας μας. Επίσης, θα ήθελα να διεξαχθούν απρόσκοπτα οι ευρωεκλογέ του 2019 και να εκλεγούν και πολλοί ε, ευρωβουλευτές με αναπηρία στο επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Thank σας ευχαριστούμε θερμά, λέει κυρία Πίγκοτ. Και σας ευχαριστώ επίσης που τηρήσατε και το χρόνο σας. Η Μαρία Πινολόπες ε, από το Ισπανικό ε, κίνημα και μέλος του ΣΕΡΜΗ, της Ισπανικής Επιτροπής Εκπροσώπων Ατόμων με Αναπηρία. Η Μαρία. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ, εκπρόσωποι των ε, κοινωνικών κινημάτων και των αναπηρικών οργανώσεων, ονομάζομαι Μαρία Πίνο. Είμαι 51 ετών, ε, προέρχομαι από την Καστίγια Λαμάντζα, μια περιφέρεια της Ισπανίας. Ε, χειραφετήθηκα χάρη στη βοήθεια των αδελφών μου. Πριν από 10 χρόνια με πήγαν σε ένα δικαστή. Έπρεπε να μιλήσω με έναν ιατροδικαστή. Με έβαλαν σε μία αίθουσα και μου άφησαν μόνη και έρημη. Κανένας δεν μου εξήγησε ε, προς τι όλη αυτή η διαδικασία. Ο δικαστής μου είπε τι θα μου αφαιρέσουν. Εγώ απλώς κουνούσα το κεφάλι μου. Έλεγα όχι, όχι. Έφυγα τρέχοντας από την αίθουσα, κλαίγοντας. Ένιωσα ανήμπορη, αδύναμη. Το 2010 ανέλαβε την κυδαιμονία μου μία οργάνωση κυδαιμονίας πλήρους ενσωμάτωσης. Παρακολούθησα μαθήματα για τα δικαιώματα που απέραν από την Σύμβαση των Ηνωμένων Αθηνών και τότε συνειδητοποίησα τι συνέβαινε. Πέρυσι έγραψα στον κυδαιμόνα μου μία επιστολή ζητώντας να αναθεωρηθεί η δικαστική απόφαση που μου αφαίρεσε τη δικαιοπρακτική ικανότητα. Πέρασα από τον γιατρό και τώρα με περιμένει δικαστήριο. Θέλω να ανακτήσω τα δικαιώματα ψήφου και χρειάζομαι βοήθεια και μόνο για τα οικονομικά ζητήματα. Μπορώ να ασκήσω αυτόνομα το δικαίωμα ψήφου. Εγώ είχα ζητήσει από τους γονείς μου παλιότερα να ψηφίσω και ψήφιζα αυτόν που ήθελα. Γιατί να μην μπορώ να ψηφίζω και τώρα. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ, θα ήθελα επ' ευκαιρία να σας ενημερώσω ότι συμμετέχω σε μια ομάδα εργασίας για την πλήρη ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία ε, και ε, συμμετέχω και στο ΣΕΡΜΗ, την Ισπανική Επιτροπή Εκπροσώπων Ατόμων με Αναπηρία. Θέλουμε να λαμβάνουμε αυτόνομα τις αποφάσεις μας, με κατάλληλη υποστήριξη. Αλλά θέλω να ακούσετε τη φωνή μας. Είμαστε κι εμείς πολίτες, ισότιμοι με εσά. Δεν είμαστε τίποτα περίεργα πλάσματα. Βοηθήστε τα άτομα με νοητική υστέρηση, με νοητική αναπηρία, με οποιαδήποτε ε, άλλη αναπηρία να μπορούν να ψηφίζουν. Στην Ισπανία 100.000 ακόμη συμπολίτε μα στερούνται του δικαιώματο ψήφου επειδή έχουν κάποια αναπηρία ή επειδή ένα δικαστή έχει αποφασίσει ότι δεν έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Μερικά άτομα έχουν νοητική υστέρηση ε, ή άλλε αναπηρίες ε, οποιασδήποτε ε, ανάπτυξης. Πάντω και στην Ισπανία, στην Ισπανική Επιτροπή Εκπροσώπων Ατόπων με, Ατόπων με Αναπηρία, δίνουμε μάχη για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Τον περασμένο Νοέμβριο η Βουλή τη Ισπανία αποφάσισε ομόφωνα να τροποποιηθεί ο εκλογικό νόμο για να κατοχυρωθεί το δικαίωμα του εκλέγην σε όλα τα άτομα με αναπηρία. Έτσι αρχίζουμε επιτέλου να σεβόμαστε και να τηρούμε και στην Ισπανία το άρθρο 29 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Το άρθρο αυτό μιλά για το δικαίωμα συμμετοχής στον πολιτικό και δημόσιο βίο των ατόμων με αναπηρία. Θέλουμε, περιμένουμε επιτέλους την άμεση μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου στην Ισπανία για να μην μεσολαβήσει καμία εκλογή στην οποία θα στερούμαστε το δικαίωμα ψήφου. Αλλά ακόμη και να ασκούμε το δικαίωμα ψήφου θα πρέπει και οι κυβερνήσεις να μεριμνούν ώστε όχι μόνο να ψηφίζουμε, αλλά να ψηφίζουμε με ισότιμους όρους με τους υπόλοιπους συμπολίτε μας. Ούτε η εκλογική διαδικασία, ούτε η προεκλογική ενημέρωση είναι προσβάσιμες για τα άτομα με δυσκολία κατανόησης. Θα πρέπει λοιπόν ε, να γίνει κατανοητή η διαδικασία, να υπάρχει προσβασιμότητα στα εκλογικά κέντρα, να ενημερώμαστε για τα πολιτικά προγράμματα, να ξέρουμε πώς θα ψηφίσουμε, θα πρέπει να δοθούν οι στοιχειώδεις πληροφορίες στα άτομα με αναπηρίες για το κοινοβουλευτικό σύστημα. Όλα αυτά θα επηρεάσουν την πρόσβασή μας στις κάλπες. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα θα ακούσουμε τον επόμενο ομιλητή, Μάρσελ Πόβλντι, από το EFHRH, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για άτομα με προβλήματα ακοής. Ευχαριστώ πολύ. Ο... Μιλάει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Ευρωπαϊκές Ελευθερίες. Σας ευχαριστώ, αλλά ως οικοδεσπότη εδώ θα ήθελα να τον παρακαλέσω τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εφαρμόσει με κεφαλαία γράμματα την προσβάσιμότητα προκειμένου να φροντίσει ότι όλες οι εκδηλώσεις όπως αυτή σήμερα να είναι και αυτές προβάσιμες για α, όλα τα άτομα με αναπηρία και να μην ε, υπάρχουν προβλήματα όπως για παράδειγμα προβλήματα υποτετλισμού που αντιμετωπίσαμε στην αρχή. Και ζητώ να σας ζητήσω την προσοχή σας για τα 52 εκατομμύρια άτομα που έχουν προβλήματα ακοής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για όλους αυτούς τους Ευρωπαίους πολίτες που θέλουν να ασκήσουν τα πλήρη δικαιώματά τους και το δικαίωμα της ψήφου και είναι απαραίτητο σε κοινοτικό, περιφερειακό και εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό ασφαλώς επίπεδο οι εκλογές να είναι προσβάσιμες με άτομα που έχουν απώλεια ακοής. Και αυτό ξεκινά με την υποτιτλισμό όλου του ενημερωτικού υλικού και του υλικού προώθησης. Επίσης όλες οι εκδηλώσεις των πολιτικών κομμάτων και άλλων των εκλογικών εκδηλώσεων θα πρέπει να είναι προσβάσιμες, να υπάρχει η σχετική πρόβλεψη και θα πρέπει να υπάρχουν διερμηνείς, ε, διερμηνείς νοηματικής στα Ολλανδικά ή, εν στη γλώσσα που μιλάει ο κάθε Και είναι δεδομένο ότι όλα τα τηλεοπτικά προγράμματα για τις εκλογικές εκδηλώσεις θα πρέπει να έχουν υποτελεσμό ανεξάρτητα από το πρόγραμμα αυτό είναι, προβάλλεται από ιδιωτικό ή από δημόσιο σταθμό. Επίσης, θα ήθελα να καλέσω σήμερα όλους τους ε, υποψηφίους όλων των πολιτικών ε, ομάδων από την αριστερά, τη δεξιά ή από το κέντρο να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις που θα είναι μόνο προσβάσιμες σε όλους. Και νομίζω ότι φέρετε πολιτική ευθύνη, κυρίες και κύριοι, και θα πρέπει να προσεγγίσετε ενώσεις που διοργανώνουν ε, εκδηλώσεις πολιτικές προσβάσιμες για όλους. Αυτό προφανώς αφορά και τους πολιτικούς υποψηφίους. Ή πρόεδρος, ε, σας ζητώ συγγνώμη, πρέπει να σας διακόψω για να σας ζητήσω να συντομεύετε παρακαλώ και να ολοκληρώσετε το συντομότερο δυνατόν. Ναι, έχω σχεδόν ολοκληρώσει. Αυτό ασφαλώς αφορά και και τους πολιτικούς υποψηφίους σε δηλεπτικά προγράμματα για την παρουσίασή τους και ε, να... να πρόκειται για προγράμματα που να έχουν πάντα υποτιτλισμό και προφανώς τα εκλογικά κέντρα θα πρέπει να είναι πάντα προσβάσιμα σε άτομα με ε, αναπηρίες και θα πρέπει επίσης και κάθε εκλογικό κέντρο να ξέρει πώς θα επικοινωνεί με τα άτομα αυτά. Θέλουμε λοιπόν τα άτομα με προβλήματα ακοής και οικοφή στην Ευρώπη να έχουν ανεξάρτητη τέτοια δικαιωμάτια ψήφου. Ευχαριστώ πολύ. Now give τώρα δίνουμε το λόγο στην πρώτη βουλευτή που θα πάρει το λόγο την Μρία Μντάλη από τη Μάλτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί φίλοι, συνάδελφοι, θα πρέπει να είμαι πολύ ειλικρινής μαζί σας. Είναι μεγάλη τιμή που βρίσκομαι εδώ σήμερα και που μοιράζομαι τις απόψεις μου μαζί σας για το τι ποιοι είναι οι λόγοι που με οδηγούν να πιστεύω ότι τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να δραματίσουν κεντρικό ρόλο στην πολιτική και δημόσια ζωή. Για μένα πρόκειται για ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με την ψηφοφορία, με το δικαίωμα ψήφου, αλλά πάει πολύ παραπέρα. Δεν πρόκειται για ένα θέμα προσβασιμότητας και μόνο, δεν πρόκειται για θέμα Πρόκειται για θέμα καθαρά ισότητος. Συνεργάζομαι στενά με άτομα με αναπηρία και με οργανώσεις αναπήρων και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στη Μάλτα τη χώρα μου. Και ένα πράγμα είναι σαφές και ξεκάθαρο. Τα άτομα με αναπηρία θέλουν ισότητα. Και είναι δικαίωμά μας να ζητούμε ισότητα όπου και να βρισκόμαστε όποιοι και αν είμαστε και βλέπω σε όλους σας άτομα τα οποία θέλουν να έχουν την ευκαιρία να κάνουν τη διαφορά. Δεν είμαστε, ε, δεν αποκλείουμε οι μεν τους δε. Είμαστε συμπληρωματικοί οι μεν προς τους δε. Και πιο σημαντικό, κανείς δεν μπορεί να καταστρώσει τέτοιε πολιτικέ για τα άτομα με αναπηρία αν δεν τι κατακτήσετε εσεί οι ίδιοι. Άρα το μήνυμά μου σήμερα είναι ένα μήνυμα ενδυνάμωση, αν θέλετε. Θα πρέπει να ακουστεί η δική σα φωνή δυνατή, ηχηρή. Δεν είναι μόνο θέμα ψήφου. Αυτό δεν νομίζω ότι εμπεριέχει την έννοια της πλήρους συμμετοχής ε, στα κοινά και στη δημόσια ζωή. Θέλω πολιτικούς υποψηφίους με αναπηρία στις εκλογικούς μας καταλόγους σε επίπεδο τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν τα κοινοβούλια μας θέλουμε πραγματικά να εκπροσωπούν όλη την κοινωνία πρέπει να αποτυπώνουν το σύνολο της κοινωνίας. Αυτό περιλαμβάνει και άτομα με πολιτική ευθύνη και με αναπηρία και τελείωσε. μου αρέσει αυτό που λέμε τίποτα χωρίς εμάς για εμάς. Μ' αρέσει αυτό το πολιτικό μήνυμα. Δεν είναι μόνο μήνυμα. Πιστεύω ότι θα πρέπει όλες οι πολιτικές να έχουν ως στόχο τους την κοινωνική συμπεριλήψη σε ό,τι αφορά και τη συμπεριλήψη ατόμων με αναπηρία για τη χάραξη πολιτικών. Ας συνεχίσουμε λοιπόν να δίνουμε δύναμη στους πολίτες μας, πολίτες μας να τους δίνουμε την ευκαιρία να κάνουν τη διαφορά. Αν είμαστε δεσμευμένοι και αν πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά και να την πετύχουμε, θα πρέπει να δώσουμε ευθύνε και δυνάμεις στα άτομα με αναπηρία και από εδώ και πέρα να δίνουμε σε όλους την δυνατότητα να είναι η φωνή τη πολιτικού γίγνεσθε προκειμένου να πετύχουμε τι αλλαγέ που επισημούμε. Ευχαριστώ πολύ και σα εύχομαι μια επικοδομητική συζήτηση. I now invite Pascal Grieb from AP. Pascal Grieb από το APF, από το Ευρωπαϊκό ε, ε, Συμβούλιο με αναπηρία ε, Nous voulons voter comme tout le monde. Θέλουμε να ψηφίζουμε όπω όλο ο κόσμο, ε, κύριε Πρόεδρε, και το δικαίωμα του εκλέγει είναι σημαντικό στοιχείο τη ιδιότητας του πολίτη και δεν είναι ένα προνόμιο που επιφυλάσσεται μόνο για λίγους παρόλα αυτά. Υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την συμμετοχή μα στα κοινά ημών των ε, ανθρώπων με αναπηρία στην και έχουμε φραγμούς ε, ε, πολλούς πρόσβαση στις πληροφορίες, στους υποψηφίους κατά την εκλογική καμπάνια. Δεν μπορούμε να πάμε στα εκλογικά κέντρα και τμήματα ε, και επίσης, επίσης υπάρχει πρόβλημα για αυτούς που ζουν υπό κυδαιμονία. Αυτά είναι κατά της Διεθνούς Συμβάσεως του ΟΗΕ. Εποτε αυτό είναι φραγμός όσον αφορά την αυτονομία μας και την ένταξή μας. Γι' αυτό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις επόμενες ευρωεκλογέ θέλει να προωθήσει το δικαίωμα και εκλέγεστε και γι' αυτό το λόγο έχουμε τις εξή συστάσεις. Πρώτα-πρώτα θα πρέπει να βελτιωθεί η προσβασιμότητα και έτσι να υπάρχει αυθεντική προσβασιμότητα και επίση θα πρέπει να, υπάρχουν, υπάρχει πολιτισμό στην επικοινωνία, να υπάρχουν κάποιοι με την ε, ε, νοματική γλώσσα και οπότε θα πρέπει να βοηθούνται και οι υποψήφοι να βγουν κάποιες ε, ενέργειες για τους ανθρώπους με αναπηρία. Επίσης να ενισχύσουμε την προώθηση στο κλινικό γίγνεσθε των αναπήρων γυναικών και αυτό να αφορά και το εκλεγή και το εκλεγήστε και στις τοπικές εκλογές και στις εθνικές και επίσης θα πρέπει αυτές οι συστάσεις να ληφθούν υπόψη ούτω ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το άρθρο 29 τη σύμβαση του ΟΗΕ. Θα πρέπει το δικαίωμα του εκλέγει και το εκλέγεστε να είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο για λίγους. Δικαίωμα για όλους. Και βαστούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που φροντίζει να υπάρχουν εγγυήσεις του δικαιώματο. Thank you very much, Pascal. Ευχαριστούμε πολύ. Πασκάλ, λέει πρόεδρος. Επόμενος ε, ομιλητής, ο Ντάνι Κανάλ, από την EUDY, Ευρωπαϊκή Ένωση των Νέων που έχουν προβλήματα ακοής. Hello everyone. I'm very... Η Ντάνη Κανάλ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τιμή μου που παρίσταμε εδώ και θα ήθελα να σας εκφράσω τις συστάσεις των ε, προσώπων του φορέα μας γιατί η επικοινωνία είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό για την άσκηση του δικαιώματος της ψήφου. Αν δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο, είναι πάρα πολύ σημαντική η σύμβαση που προβλέπει ότι θα πρέπει να έχουν προσβασιμότητα και αυτοί που έχουν προβλήματα ακοής. Αλλά βέβαια θα πρέπει πρώτα πρώτα να εντάσσονται όλοι στη διαδικασία του εκλέγην γιατί θα πρέπει να υπάρχει νοηματική γλώσσα που να εξηγεί τα σχετικά και σύμβολα. Άρα χρειάζεται αυτού του είδους η επικοινωνία, κάτι το οποίο δεν ισχύει σήμερα και θα, έτσι θα πρέπει να χορηγούνται οι κατάλληλες πληροφορίες. Σήμερα επομένω, δεν έχουμε δικαίωμα ε, στο εκλέγγυ γιατί δεν ε, υπάρχει μετάφραση σε νοηματική γλώσσα και έτσι οι νέοι οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική ε, υφίστανται αυτού του είδους τον αποκλεισμό που είναι διπλώς, γιατί έχουν αναπηρία. Θα πρέπει ομένως οι άνθρωποι με αναπηρία να αποκτήσουν το δικαίωμα στο εκλέγην. Ε, αυτό θα πρέπει να κάνουμε, να υπάρχει ισότητα όσον αφορά την πρόσβαση στην ψηφοφορία. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ την ε, Ντάνη για τώρα. Ο τελευταίο από τον κατάλογο των ομιλητών που έχω εγώ είναι ο Τζούλιο Ναρντόνα και κατόπιν θα πάρει τη σκητάλη άλλο για να προεδρεύσει από το Ιταλικό Φόρμιο του ανθρώπου με αναπηρία. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εμείς υπογράφουμε αυτό το κείμενο που από το Ιταλικό Φόρουμ για τα πρόσωπα με αναπηρία θέλουμε να μπορέσουν όλοι όσοι έχουν αναπηρία να ψηφίζουν αυτόνομα. Δεδομένου ότι το άρθρο 9 της Συμβαστορίας του τα δικαιώματα των προσώπων με αναπηρία ε, ορίζει ότι όλα αυτά τα πρόσωπα θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να πάνε σε ιδιωτικά ή κρατικά κτίρια και, και στο ίντερνετ όπως όλοι οι άλλοι. Επειδή σήμερα το Διεθνές Σύμβολο για την προσβασιμότητα είναι ε, αναπηρική καρέκλα και κάθε μέρα έχουμε τέτοιου είδους ε, τέτοιους παραστάσεις στη θεμενή ζωή ε, όσον αφορά την ελευθερία της διακίνησης ενός προσωπού που χρησιμοποιεί αναπηρική καρέκλα και αυτή όμως είναι εσφαλμένη εντύπωση όμως είναι διαδεδομένη αλλά έχει φτάσει στις δημόσιες αρχές και στα μέσα ενημέρωσης. Οπότε θα πρέπει αυτοί οι φραγμοί να αρθούν και θα πρέπει επομένως να υπάρχουν οι κατάλληλε παραστάσεις, οδηγίες για προσανατολισμό και ασφάλεια όσων έχουν προβλήμα με τις αισθήσει τους. Γι' αυτό και εμείς που προσυπογράφουμε ε, αυτό το, το αίτημα ε, καλούμε το EDF ούτως ώστε να προωθήσει μια ε, πρόταση για να χρησιμοποιείται αυτό το διεθνές σύμβολο. Να υπάρχουν και άλλες γραφικές ε, παραστάσεις και ενδείξεις ούτως ώστε να αντιμετωπίζονται οι διάφορες καταστάσεις δυσχέρειας αυτών των προσώπων ακόμη και όταν δεν εμπίπτουν στην αναπηρία Χρειάζεται μέρος να υπάρχει με συγκεκριμένο αυθεντικό τρόπο προσβασιμότητα και αυτό προσπάθησε να κάνει ε, η εταιρεία των Ιταλικών σιροδρομων για ένα τέτοιο ε, σύμβολο. Να, αυτό σας το προτείνουμε ως μια πιθανή λύση. Σας ευχαριστούμε, λέει κυρία Πίγκοτ. Ευχαριστούμε Τζούλιο και για τις πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις σου. Ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους που έλαβαν το λόγο σε αυτό το πρώτο τμήμα της συζήτησης και τους ευχαριστώ θερμά που τήρησαν και το χρόνο αγόρευσης. Δίνω το λόγο στον Άνταμ Κώσσα που φαντάζομαι θα είναι πολύ καλύτερο συντονιστής ε, της συζήτησης από ότι εγώ. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Άνταμ Κώσα. Ευχαριστώ, κυρία Πίγκοτ. Όχι, πραγματικά ήταν ε, θαυμάσια η δική σου προσπάθεια. Συντόνισες ε, επάξια το πρώτο τμήμα της συζήτησης. Ε, θα ήθελα και εγώ να απευθύνω μια θερμή παράκληση. Έχετε μπροστά σας μια μικρή οθόνη. Ε, στα τραπέζια μπροστά σας στα έδρανα. Εκεί υπάρχει και χρονόμετρο. Ρίχνετε μια ματιά για να βλέπετε πόσος χρόνος έχει απομείνει και να μην το ξεπερνάτε. Θα δώσω τώρα το λόγο στον συνάδελφο Ευρωβουλευτή, τον κύριο Μπενιφέη. Σήμερα είναι εξαιρετική αυτή η περίσταση και μεγάλη μας χαρά βρισκόμαστε εδώ για να αποδείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να φροντίσει για εσάς ώστε όλα να βελτιωθούν γιατί ακόμα δεν έχουμε φροντίσει να παράσχουμε εγγυήσεις πλαισίωσης των προσώπων με αναπηρία. Θα πρέπει να υπάρχει προσβασιμότητα, θα πρέπει να υπάρχει κάποια συνοχή και όπως σωστά τα είπαν όσοι μίλησαν πριν από μένα, Κάτι γνώμη μου θα πρέπει σήμερα να προβάλλουμε αυτό το δικαίωμα στην προσβασιμότητα, θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προβεί σε διαπραγματεύσουν τα κράτη-μέλη. Δεν είναι δυνατόν να δεχόμαστε ε, εκπτώσεις από τέτοια δικαιώματα. Δεν είναι δυνατόν να ωφελούνται οι λίγοι με τέτοιου είδους ε, απεμπόληση δικαιωμάτων. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει συμμετοχή στα κοινά, στα πολιτικά. Και αλλιώς η ίδια η δημοκρατία πάσχει να συμμετάσχουν αυτοί που έχουν αναπηρία. Σας ευχαριστούμε ε, γιατί με τις προσπάθειές σας μας βοηθήσατε ως νομοθέτες. Ευχαριστούμε όλους όσους ήρθαν εδώ και τους συναδέλφους, ε, τους συμπολίτε μας, τους Ιταλούς, και όλους που έχουν συμμετάσχει σε αυτό γιατί ακριβώς τίποτα που σας αφορά δεν θα γίνει χωρίς την ε, ε, συμμετοχή σας. Χίλια ευχαριστούμε. Ο κύριος Κώσα. Σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στην επόμενη ομιλητριά μας, την κυρία Άννα Χίλντινγκσον, από την Σουηδική Ομοσπονδία Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία. Παρακαλώ, κυρία Χίλτβινσον, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το 1989 ε, άτομα με νοητική αναπηρία επέκτησαν το δικαίωμα ψήφου στη Σουηδία. Επιτέλους ε, γίναμε κι εμείς ε, ισότιμοι πολίτες, πλήρεις πολίτες. Ε, αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό. Δεν μπορούμε να έχουμε στην ίδια χώρα πολίτες δύο, κατηγορία, δύο κατηγοριών. Δηλαδή, ε, πολίτες πρώτης κατηγορίας με δικαίωμα ψήφου και πολίτες δεύτερης κατηγορίας ε, που δεν έχουν ικανότητα ψήφου. Βέβαια, η νομική, η νομοθετική κατοχήρωση του δικαιώματος ψήφου είναι απλώς το πρώτο βήμα. Γιατί το χρόνο που ακολούθησε από την επίσημη έγκριση της νομοθεσίας που κατοχύρωσε αυτό το δικαίωμα ψήφου μέχρι την πραγματική συμμετοχή στις εκλογές των ατόμων με αναπηρία πέρασε πολύ καιρό. Το θέμα ε, δεν είναι απλώς να πάμε να ψηφίζουμε, αλλά να έχουμε εκ των προτέρων καλή ενημέρωση ώστε να μπορούμε να ψηφίζουμε εμπεριστατωμένα. Όλο και περισσότερο πάντως τα άτομα με αναπηρία ασκούν το δικαίωμα ψήφου τους και στην Σουηδία. Και είναι φυσικό γιατί οι πολιτικές αποφάσεις επηρεάζουν την καθημερινότητά τους. Μάλιστα συμμετείχαμε σε ένα πρόγραμμα ε, που έδινε την ευκαιρία στα άτομα με αναπηρία να μαθαίνουν πώς λειτουργεί η κοινωνία. Και μάλιστα οι περισσότεροι από αυτούς που παρακολούθησαν αυτή την κατάρτιση κατάφεραν και άσκησαν το δικαίωμα ψήφου τους στις επόμενες εκλογές. Η γνώση σημαίνει δύναμη, σημαίνει εξουσία και θα, δεν θα πρέπει κανένα άτομο με αναπηρία να στερείται του δικαιώματος ψήφου. Επίσης θα πρέπει να προηγείται πρόσβαση σε εύληπτες κατανοητές πληροφορίες. Αυτό είναι απαραίτητο. Επίσης, ε, ε, τα μέτρα που είναι ε, απαραίτητα για λίγους είναι καλά και για τους πολλούς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει ο κύριος Κώσα. Και σε ευχαριστούμε, Άννα, που τήρησες και το χρόνο μιλία σου. Θα δώσω τώρα το λόγο σε μια συνάδελφο ευρωβουλευτή από τη Σλοβακία, την κυρία Γιάννα Ζητνάσκα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο, κυρία Ζητνάσκα. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητές κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή για μένα που βρίσκομαι εδώ μαζί σας σήμερα και επιτρέψτε μου ιδιαίτερως ε, να καλωσορίσω τη Σλοβακική αντιπροσωπεία και χαίρομαι ιδιαίτερως ε, που ήρθατε τόσο πολύ άρθιμοι. Είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουν στην πολιτική ζωή και άτομα με προβλήματα υγείας. Στο πνεύμα της δημοκρατίας ε, προασπίζεστε και αγωνίζεστε για τα δικαιώματά σας, τα δικαιώματα των παιδιών σας, των παιδιών σας, των ε, συντρόφων σας. Ε. Αλλά ένα σημαντική, μια σημαντική προϋπόθεση για τη χάραξη της πολιτικής είναι να συμμετέχει κανείς στην χάραξη της πολιτικής αυτής. Άρα διαπιστώνουμε ότι τα άτομα με αναπηρία σε πολλές περιπτώσεις ε, ε, ούτε να ψηφίσουν ούτε να κατέβουν υποψήφοι μπορούν. Και Αυτό αφορά σε πολλές περιπτώσεις και ακραία φαινόμενα που παρουσιάζονται στην πολιτική ζωή. Χτες ε, είχαμε μία εκδήλωση για το θέμα της Βερόνικα Χαμηλετότουμα από τη Σλοβακία σε ό,τι αφορά την κράτηση της σε στρατοπέδας συγκέντρωσης ε, στην. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, τα άτομα με αναπηρία και με διανοητική αναπηρία ήταν ε, στο στόχο του ναζιστικού καθεστώτος που πρέβησε σε μαζικές ε, εκτελέσεις. Αυτό το ρεπορτάζ ε, διατίθεται και στο διαδίκτυο με αγγλικούς υπότιτλους. Ε, αν θέλετε προφανώς μπορείτε να μας ζητήσετε και να σας ε, δώσουμε περισσότερες πληροφορίες. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω και άλλη μια παρατηρήση. Αυτό το φρικτό παρελθόν δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε να συνεχιστεί. Θα πρέπει μαζί λοιπόν να τα καταφέρουμε και πιστεύω ότι μπορούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στον επόμενο μελητή από τη Λιθουανία, τον Βιλάλ Κάιτε. Έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω σε αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση. Θα μιλήσω εξ ονόματα ε, του Ευρωπαϊκού Φόρουμ, του Λιθουανικού Φόρουμ για την με αναπηρία. Αντιμετωπίζουμε νομικά προβλήματα στη Λιθουανία, προβλήματα προσβασιμότητα και προβλήματα στάσης σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή μας στην πολιτική ζωή. Το 2016 έγινε γενικές εκλογές και 60% των εκλογικών κέντρων δεν ήταν διαμορφωμένα σύμφωνα με τι ανάγκε των ατόμων αναπηρία. Κατά τη διάρκεια της προεκλογική εκστρατεία, όλο το εκλογικό υλικό δεν ήταν προσαρμοσμένο. Οι πληροφορίε ευανάγνωστε, δεν διατέθηκαν, δεν ήταν σωστή ποιότητα. Τα άτομα, οι τύφλοι δεν μπορούσαν να ψηφίσουν μόνοι του, ανεξάρτητα. Και δυνατότητα να ψηφίσει κανείς από το σπίτι δεν συνεπάγεται η αντιμετώπιση, συμπερίληψη και συμμετοχή. Τα άτομα με διανοητική αναπηρία αντιμετωπίζουν διακριτική μεταχείριση γιατί κηρύσσονται ε, νομική ανικανότητα και ο νόμος δεν επιτρέπει στα άτομα αυτά να ψηφίσουν. Διαγράφονται από τους εκλογικούς καταλόγους και αυτή η δικαιοπρακτική πρακτική ικανότητα αφορά πολλούς τομείς της ζωής. Η έλλειψη αυτή νομική ικανότητα και σε ό,τι αφορά την άσκηση τέτοιων δικαιωμάτων όπω το δικαίωμα τη ψήφου. Τέτοιε λοιπόν αποφάσει λαμβάνονται μόνο βάσει ιατρικών κριτηρίων. Αυτό λοιπόν παραβιάζει τα δικαιώματα των πολιτών σε ό,τι αφορά την συμμετοχή στα κοινά της χώρας. Το άρθρο 29 της Σύμβασης μιλάει για τα ίσα δικαιώματα για τα άτομα με αναπηρία και την ισότητα που απολαμβάνουν όλοι ενώπιον του νόμου. Αυτό θα πρέπει να κατοχυρώνεται αν θέλουμε τέτοια άτομα να αποτελούν τμήμα της κοινωνικής και της πολιτικής μας ζωής. Η κοινωνία μας θα πρέπει να βασίσει τη στάση της ε, στο γεγονός ότι είναι αναπαλουτρίωτο το δικαίωμα των ανθρώπων αυτών να συμμετέχουν στην πολιτική και κοινωνική ζωή. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο στο Βελγικό Φόρουμ για πρόσωπα με αναπηρία στον κύριο Ζουλιάν Ποστιό. Καλημέρα, ονομάζομαι Ζουλιάν Ποστιό. Είμαι ο πρόεδρος του φορέα του ΕΝΟ, περιοχής του Βελγίου, για την αυτοεκπροπόρηση. Έχουμε διανοητικές ε, δυσκολίες, έχουμε διανοητική αναπηρία και εκπροσωπούμαστε στο BDF το Βελγικό Φόρουμ. Εκεί που προσωπούνται τα πρόσωπα με αναπηρία που διεκδικούν συμμετοχή στο πολιτικό γίγνεσθε. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε υποχρεώσεις και δικαιώματα και δεν σας ε, να σας πω για τις εκλογές, να σας πω την εμπειρία μου όσον αφορά τις εκλογές. Την πρώτη φορά που πήγα να ψηφίσω δεν ήξερα ποιον υποψήφιο να διαλέξω και ψήφισα ό,τι ψήφισαν και οι γονείς μου και δεν μπορούσα να διαμορφώσω κάποια γνώμη δεν μπορούσα να ταυτιστώ με κάποιο προεκλογικό πρόγραμμα οπότε αυτά που λέγανε υποψήφοι δεν τα καταλάβαινα είχα φίλους που δεν μπορούσαν ούτε να διαβάσουν ούτε να γράψουν άρα δεν μπορούσαν να ασκήσουν το δικαίωμά τους και θα μπορούσαν να γίνουν διάφορα. Θα πρέπει τα προγράμματα των υποψηφίων να είναι ευανάγνωστα, να είναι κατανοητά. Αυτό θα ωφελήσει όλους. Θα πρέπει να μπορούμε να ασκήσουμε τα δικαιώματα μας και να είμαστε υπεύθυνοι πολίτες. Αυτό είναι το σωστό για την κοινωνία. Οπότε και αν μπορέσετε να μας βοηθήσετε ε, και εμείς θα είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε και καλημέρα σας. Köszönöm, kiválóan betartotta az Σας ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε που τηρείτε τα χρονικά όρια. Μπράβο σας. Και τώρα να δώσουμε τον λόγο σε έναν συνάδελφο ευρωβουλευτή, τον Λουίτζι μοργκανο Πρώτα πρώτα εσάς να ευχαριστήσουμε που ήρθατε εδώ και σας το λέω γιατί εδώ μπορούμε να κάνουμε κάτι για το μέλλον αλλά και για το παρόν. Το προήμιο του χάρτη Ευρωπαϊκών Γεμάτων λέει ότι οι λαοί της Ευρώπης, Ευρώπης φτιάξαν αυτή την Ευρώπη και θέλουν να βασίζεται σε κοινέ αξίες. Θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι έχουμε κοινή πνευματική πολιτική κληρονομία και έχουμε αυτές τις παγκόσμιες αξίες της αξιοπρέπειας, της ισότητας, της αλληλεγγύης και βασίζεται η Ένωση, έχει θεμέλιο την δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Και στο επίκεντρο όλων είναι ο άνθρωπος, η ιδιότητα του πολίτη και έτσι θα έχουμε έναν χώρο ελευθερίας, δικαιοσύνη και δημοκρατίας. Και επομένω είναι αυτονόητο, όπως ορίζει και το άρθρο 29 της ε, Σύμβασης, ότι δεν απαγορεύεται πάσα δυσμενής διάκριση. Και επομένω, θα πρέπει όλες αυτές οι αρχές να υλοποιούνται και να μπορούν οι άνθρωποι με αναπηρία να απολάβουν των δικαιωμάτων τους σε όλα τα δικαιώματα της ε, κίνησης, διακίνησης, της ελευθερίας έκφρασης και φυσικά στο δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεστε. Και θα πρέπει βέβαια να υπάρχει η σχετική στρατηγική. Τα ξέρει η κυρία Στίβενς που κάθεται εδώ. Οπότε και το Κοινοβούλιο απευθύνθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είπαμε θα πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικές ρυθμίσεις για την προσβασιμότητα στους δημόσιους χώρους και θα πρέπει ενδεχομένως να εγκρίνουμε την πρόταση του εκπροσώπου του Ιταλικού Φόρουμ του Κιλίου Ναρντόνε να υπάρχουν δηλαδή επιπλέον ενδείξεις και σήματα σε κάθε χώρο για κάθε είδους δυσκολία και αναπηρία ό,τι επιδέχεται διευκόλυνση και λύση. Καλή πτυχία στις εργασίες μας. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα έχουμε άλλον εξέχοντα ε, συνάδελφο, από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κυρία λάρα Κόμη. Καλώς ορίσατε όλοι. Θερμά σας αγκαλιάζουμε, σας φιλούμε, μια που σήμερα δίνετε ένα παράδειγμα για μας. Ε, αυτό που κάνετε είναι ενθάρρυνση ε, για την καθημερινή δουλειά μας. Και αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να πέσουν όλοι οι φραγμοί, να αρθούν όλες τις μενείς διακρίσεις όσα Κάθε μέρα σας δυσκολεύουν στην ε, ζωή σας. Εδώ να νιώθετε σας στο σπίτι σας, γιατί εμείς ε, εκλεγήκαμε για να σας εκπροσωπούμε. Πολύ σωστά λέμε για καλύτερη προσβασιμότητα στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος. Πάντως να σας πω ότι το 2019 θα ήθελα να σας δω εδώ ως ευρωβουλευτές. Να μην είμαστε μόνο παθητικοί ψηφοφόροι, αλλά ενεργοί μπορείτε, πρέπει να είσαστε εσείς να γίνετε ε, εδώ εκπρόσωποι στα θεσμικά όργανα και βεβαίω να σε ευχηθώ καλές ε, γιορτές ε, και κάθε ευτυχία γιατί έχετε δικαίωμα στην ευτυχία να μπορέσετε να κάνετε ό,τι θέλετε εσείς και η οικογένειά σας ποτέ δεν σας ξεχνούμε, σας θεωρούμε ότι είσαστε και εσείς όπως όλοι οι άλλοι δεν είστε μόνοι. Ναι στην πολιτική εκπροσώπηση, αλλά ε, πρώτα πρώτα να είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε ε, συνάδελφοι. Είμαστε στο πλάι σας και σας βοηθούμε, σας υποστηρίζουμε. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Κόμη και τώρα. Εδώ ολοκληρώνω την δική μου προεδρία και δίνω την σκητάλη στον συνάδελφο τον κύριο Πλούρα. Αλλά πρώτα πρώτα θέλω να σας πω το εξής που μας αφορά όλους. ότι εσείς συμμορφώνεστε πολύ περισσότερο και προσαρμόζεστε πολύ καλύτερα στο χρονικό όριο των αγορεύσεων από ότι οι συνάδελφοί μου ευρωβουλευτέ. Να, που μας δίνετε ένα παράδειγμα προς μίμηση. Πρέπει να κάνουμε και εμείς όπως εσείς. Κύριε Πλούρα, έχετε την σκητάλη της Προεδρίας. Σε ευχαριστούμε, Άντα. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Ρούντολφ Βολέινικ, που είναι αντιπρόεδρος της ενοποιημένης οργάνωσης των τυφλών και χόντων προβλημάτων όρασης της Τσεχίας. Παρακαλώ, κύριε Βολέινικ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ε, κυρίες και κύριοι αξιότιμοι συνάδελφοι, είμαι ε, αντιπρόεδρος της ε, αντιπροσωπευτικής οργάνωσης των τυφλών και των εχόντων προβλημάτων όρασης με βάση τα κριτήρια που θεσπίζονται στην Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Ε, η οργάνωσή μας ε, δεν είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου των Ατόμων με Αναπηρία για λόγους που ε, είναι εκτός θέματος για τη σημερινή εκδήλωση. Θα ήθελα πάντως να σταθώ εν συντομία σε δύο θέματα που περιλαμβάνονται στο μανιφέστο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ των Ατόμων με Αναπηρία. Καταρχήν, σε οποιαδήποτε ψηφοφορία οι τυφλοί θα έχουν πρόβλημα προσβασιμότητας στο μέτρο που η διαδικασία στηρίζεται μόνο σε τυπωμένα φυλάδια και ψηφοδέλτια. Γιατί ε, τη στιγμή που ε, χρησιμο, α, με ηλεκτρονικά 0 και 1 το έντυπο υλικό μπορεί εύκολα να αποτυπώνεται σε μπράγια, σε μεγαλύτερα, μεγαλύτερους χαρακτήρες ή με, ε, να φαίνεται με άλλη μορφή ώστε να μπορούν και οι τυφλοί με απόλυτη ε, απομόνωση και αυτονομία να ψηφίζουν. Είναι απλούστατη η αλλαγή της διαδικασίας. Δεύτερο θέμα αφορά την ψηφοφορία για τα άτομα με αναπηρίες που μέχρι στιγμής ε, δεν μπορούσαν να ψηφίσουν. Υπό την επιφύλαξη λοιπόν των δικαιωμάτων αυτών των ατόμων θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε να αποτρέψουμε τους λαοπλάνους, τους λαϊκιστές στην καλύτερη περίπτωση, τους ε, ακραίους ε, στη χειρότερη περίπτωση, να τους αποτρέψουμε από την ψηφοθυρία θα ήθελα εν κατακλείδη να ευχαριστήσω την Ευρωβουλευτήνα Όλγα Σεχνάλοβα που είχε την καλοσύνη να μας προσκαλέσει σε αυτό το τέταρτο Ευρωκοινοβούλιο των ατόμων με αναπηρία. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστούμε, λέει ο κύριος Πλούρα. Και τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Βέρα Μπομβαλό από την Πορτογαλική Οργάνωση BIF. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ. Είμαι η Βέρα Μπομβαλό και εκπροσωπώ το ε, Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναφύριες για όσους έχουν ε, εγκεφαλικές ε, κακώσεις και κάποια εγκεφαλική αναπηρία πολύ... Ε, κάποιος που έχει υποστεί μια εγκεφαλική κάκωση ε, γίνεται άλλος άνθρωπος, ε, δεν έχει συγκέντρωση, χάνει τη μνήμη του, έχει περίεργη συμπεριφορά. υπάρχουν δύο κόσμοι για αυτόν τον άνθρωπο. Ο προηγούμενος κόσμος της ζωής του, στον οποίο ήταν ελεύθερος να συμμετέχει, και ο νέος κόσμος που είναι ο κόσμος μετά την αναπηρία του εκεί πειράζεται η απασχόληση, η μεταφορά. Μερικές φορές αυτή η τομή είναι απρόσιτη πια για τον τραυματία και όσοι έχουν τέτοιες ε, νευρολογικές σοβαρές ασθένειες ε, είναι, μένουν εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους, δεν έχουν δυνατότητα επικοινωνίας, ε, κινητικότητας, δεν μπορούν να συμμετέχουν στον ενεργό βίο, δεν μπορούν να ψηφίζουν. Είμαστε στο 2017 και με, έχουμε ακούσει πολλά λόγια για αξίες, για καινοτομία, για ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτές όμως οι αποφάσεις δεν αγγίζουν όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, ιδιαίτερα αυτούς που έχουν μια αναπηρία, ορατή ή άδειλη. Γιατί ε, δεν είναι το θέμα της νοοτροπίας που έχει πρόβλημα λείπει η πολιτική βούληση, γιατί όλοι είμαστε ε, δυνητικά ανάπηροι, με οποιαδήποτε αναπηρία. Θα πρέπει λοιπόν οι αποφάσεις μας να καλύπτουν όλες τις πιθανότητες αναπηρίας. Και σας παρακαλώ, στο έργο σας το καθημερινό, δώστε προτεραιότητα στην αναπηρία και λάβετε την υπόψη σε κάθε τομέα εργασία και απόφαση. Ε, θα ήθελα να πω στους παρόντες ευρωβουλευτές, αλλά κυρίως τους απόντες, να φροντίσουν ώστε να μην υπάρχουν δύο διαφορετικοί κόσμοι. Θα ήθελε η Ευρώπη να είναι ένας χώρος για όλους τους πολίτες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, λέει, λέει ο κύριος Πλούρα. Και περνάμε στον κύριο Όσβαλτ Φέλερερ από το κέντρο ε, αυτόνομης λήψης αποφάσεων για τους ε, ανθρώπους με αναπηρία από την Αυστρία. Hello. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αγαπητοί ευρωβουλευτές και εκπρόσωποι, ονομάζομαι Όσταρτ Μπολέτ και χαίρομαι ιδιαίτερος που μπορεί παρό... να βρίσκομαι εδώ και να μιλία γερμανικά. Το κέντρο αυτόνομης ε, λήψης αποφάσεων στην Βιέννη διακηρύσει ότι ο καθένας είναι αυτόνομος και ότι όταν είναι κανείς αυτόνομος δεν πρέπει να προσέχει τι λέει. Είμαστε ένωση υπόδεγμα για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει η αυτόνομη λήψη αποφάσεων αποφάσεων. Στο κέντρο λοιπόν στην Βιέννη θέλουμε ίσα δικαιώματα με άτομα με μαθητικές δυσκολίες γιατί τα άτομα με τέτοιες δυσκολίες θα πρέπει σίγουρα να εκπροσωπούνται στην πολιτική ζωή. Και έχουμε και στο σχετικό άρθρο αναφορά στο άρθρο 29. Και η δικτύωση με άλλες οργανώσεις ε, αυτόνομης λήψη αποφάσεων είναι επίσης πολύ σημαντική, γιατί από κοινού μπορούμε να, να πετύχουμε πιο πολλά. Αυτή η δικτύωση λοιπόν παίζει σημαντικό ρόλο. Και γι' αυτό λοιπόν βοηθά και η ανταλλαγή απόψεων εδώ σήμερα και η ενίσχυση όλων μας. Τέτοιες εκδηλώσεις θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα πιο συχνά. Για την βοήθεια πιο πολλών ανθρώπων, πολλά άτομα με Εκπαιδευτικέ και μαθητικές δυσκολίε δεν έχουν την δυνατότητα, δεν έχουν οικονομικά μέσα για να έρχονται σε τέτοιες εκδηλώσεις, εκδήλωσεις. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ σήμερα και προσβλέπω στις επόμενες ημέρες ε, τίποτα για εμάς χωρίς εμάς. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Μπρενσλάφ Μαμόικα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναπηρίας. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να μιλήσω για την ιδιαίτερη σημασία και για την αποτελεσματικότητα των οργανώσεων για άτομα με αναπηρία. Τα δικαιώματα των πολιτών με αναπηρία είναι σημαντικά και για αυτούς λοιπόν ο διάλογος αυτός παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Εκτός αυτού θα ήθελα να τονίσω ένα ιδιαίτερο μέτρο, την οδηγία για την προσβασιμότητα των κτηρίων δημόσιας δίκησης. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ε, μεγαλύτερη προσβασιμότητα της δημόσιας ζωής και σε ό,τι αφορά το θέμα της ψήφου για τα άτομα με αναπηρία. Η οδηγία αυτή αναφέρει και το θέμα της υποψηφιότητας και των ανεξάρτητων υποψηφίων. Για παράδειγμα και οι φοιτητέ δεν έχουν δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες αυτές. Τίθεται θέμα, για παράδειγμα, σπουδών, αν μπορεί να σπουδάσει κανείς. Γι' αυτό, λοιπόν, θα ήθελα να σας παρακαλέσω, άξιοτιμοι βουλευτές, να συμμετάσχετε ενεργά στον διάλογο με τις οργανώσεις μας προκειμένου να μπουν περαιτέρω διατάξεις στην ομοθεσία που θα τονίσουν την, ε, το ρόλο μας. Σας ευχαριστώ και τώρα ο λόγος στον κύριο Γιάν Φίλιπ Λιμπίτσκι που είναι μέλος της Πολωνικής Γερουσίας. Κύριε Γερουσιαστά, έχετε το λόγο. Παρακαλώ, ανοίξτε το μικρόφωνο σας. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, είμαι γερουσιαστής από την Πολωνία, άτομα με αναπηρία και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας για τα άτομα με αναπηρία στην Πολωνική Βουλή. Θα ήθελα να πω καθαρά και εξάστερα ότι οι Πολωνοί πολίτες με αναπηρία θέλουν να λαμβάνουν μέρος στις εκλογές, ε, μεταξύ άλλων, γιατί ε, εκεί που υπάρχουν περισσότερα άτομα με αναπηρίες ε, διαμορφώνονται και με ιδιαίτερο τρόπο τα εκλογικά κέντρα. Και στην κοινοβουλευτική θητεία που ολοκληρώθηκε το 2015, εισαγάγαμε στην Πολωνία διευκολύνσεις ε, για τη συμμετοχή στις εκλογές των ατόμων με αναπηρία. Υπήρχε δυνατότητα ψηφοφορία, της ψήφου με λιλογραφία ή μέσω πληρεξουσίου. Επίσης υπήρχε δυνατότητα χρήσης ειδικών ε, ε, μέσων ε, για άτομα με προβλήματα όρασης ή τυφλούς. Επίσης, έχουμε προβλέψει και τη δυνατότητα ψηφοφορίας μέσω του διαδικτύου. Δυστυχώς όμως, το τελευταίο καιρό προτάθηκε ένα νομοσχέδιο από τη νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία που περιορίζει πολλά τέτοια δικαιώματα. Ο, καταργεί το δικαίωμα ψήφου με αλληλογραφία. Ε, για αυτή την επιδείνωση σας έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου προηγουμένως ο κύριος Πλούρα. Επίσης, ε, έτσι θα νοθευτεί το ε, αποτέλεσμα ή το, επιχείρημα που χρησιμοποίησε η κυβέρνηση για την κατάργηση του ψήφου διαλογραφίας. Διαμαρτύρομαι εντόνως. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και δεν νομίζω ότι οι Πολωνοί ε, ψηφοφόροι με αναπηρία δημιουργούν απειλή για τη σωστή διεξαγωγή των εκλογών ή απειλούν με νόθευση τις εκλογές. Και η απειλή της ε, εκλογικής νοθείας ε, νομίζω είναι ένα ψεύτικο επιχείρημα που χρησιμοποιεί η πολωνική κυβέρνηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ευρωβουλευτή Μάρεκ Πλούρα για την πρόσκληση και για το ότι μου έδωσε την ευκαιρία να λάβω το λόγο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκ μέρους ε, πολιτών που έχουν κάποια αναπηρία. Ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Γερουσιαστά και όντως ε, συμφωνώ ότι ήδη στη χώρα μας απολαμβάνουμε κάποια πράγματα που ε, ακόμη μερικοί Ευρωπαίοι μόνο ονειρεύονται. Ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Κοζουόφ Καραγεύητς. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους προτεργάτες και τους διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης του τέταρτου Ευρωκοινοβουλίου των ατόμων με αναπηρία έτσι κάνουμε μια αξιολόγηση των μέχρι τώρα πρόοδων και επιτευγμάτων και διαπιστώνουμε τι προκλήσεις έχουμε ακόμη να αντιμετωπίσουμε μέχρι ότου εξασφαλίσουμε την ισότιμη ε, αντιμετώπιση όλων των πολιτών. Ευχαριστήσω την κυρία Στίβενς, τον κύριο Κώστα, τον κύριο Πλούρα που είναι η Αγία Τριάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι οι φύλακες άγγελοι των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία γιατί η άνηση μεταχείριση, οι διακρίσεις ε, είναι κάτι που δεν συνάδει με τις θεμελιώδεις αρχές, αλλά ούτε και με αρχές των ε, ε, κρατών μελών. Γιατί η ισότιμη αναγνώριση προϋποθέτει συμμετοχή και στις εκλογές και συμμετοχή στην χάραξη αποφάσεων και συμμετοχή στον πολιτικό βίο και των ατόμων με αναπηρία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και το επισημάναμε επανειλημμένο σήμερα. Και μάλιστα ε, τα δικαιώματα αυτά δεν θα πρέπει απλώς να κατοχυρώνονται στη θεωρία, στα χαρτιά, αλλά να εφαρμόζονται και στην πράξη. Θα πρέπει και για τις εκλογές να καταργήσουμε τα εμπόδια. Είμαστε στο 2017 και μας βοηθάει η τεχνολογία. Χάρη στην τεχνολογία μπορούμε να καταρρύψουμε τα εμπόδια και τους φραγμούς και μάλιστα με πολύ πιο φθηνό τρόπο. Το θέμα δεν είναι πια οικονομικό, το θέμα είναι πια πολιτικό. Χρειάζεται πολιτική βούληση. Τα τελευταία χρόνια η Πολωνία έχει εισάγει κάποιες ρυθμίσεις που διευκολύνει τους, ε, ε, τα άτομα με αναπηρία να συμμετέχουν στις εκλογές κάθε επίπεδο ε, και στις δημοτικές. Επίσης υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής ή ψηφοφορίας διαλληλογραφίας μέσω πληρεξουσίου και ούτω καθεξής. Βέβαια, τελευταία έχει υποβληθεί ένα νομοσχέδιο που καταργεί κάποια τέτοια δικαιώματα. Ελπίζω να ξέρουν οι βουλευτές πώς θα σταθούν απέναντι σε αυτή την ψηφοφορία άσχετα με την πολιτική τους παράταξη και θα λάβουν υπόψη τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Ε, και για αυτά τα θέματα, για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία, είναι προς όφελος όλων μας η πρόοδος και όχι η παλινδρόμηση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία λέει ο κύριο Πλούρα. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Τουπιλούση Τουντορέλ, που εκπροσωπεί το Ρουμανικό Εθνικό Συμβούλιο των Ατόμων με Αναπηρία. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί Ευρωβουλευτέ, κυρίες και κύριοι, λέγομαι του Τουντορέλ. του Ντορέλ, εκπροσωπώ το Ρουμανικό Εθνικό Συμβούλιο Ατόμων με Αναπηρία, το CNDA. E. Θα ήθελα εκ μέρους οργάνωσής μας να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την εξαιρετική εκδήλωση και να ευχαριστήσω την κυρία Νόριτσα Νικολάη, την Ευρωβουλευτή που ε, μας προσκάλεσε και χάρη στην οποία βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα και αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι μια ένωση ίσων πολιτών από όποια χώρα και αν κατάγονται, σε όποια κατάσταση και αν βρίσκονται, αν έχουν αναπηρία ή όχι. Η Ευρώπη θα πρέπει να μας επιτρέψει να υλοποιήσουμε τα όνειρά μας και να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το δυναμικό μας. Και γι' αυτό δεν θα πρέπει να αποκλείουμε από τη συμμετοχή σε αυτή την Ευρώπη τα άτομα με αναπηρία. Θα, πρέπει να τους επιτρέπουμε τη συμμετοχή στο πολιτικό βίο και την άσκηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων. Γι' αυτό και προτείνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την υιοθέτηση μιας οδηγίας που θα επιτρέπει στα άτομα με αναπηρίες την απόλαυση ίσων δικαιωμάτων με αυτά που απολαμβάνουν οι εθνοτικές μειονότητες. Δηλαδή θα πρέπει να έχουν εκπροσώπους ε, στις νομοθετικές ε, δομές και στα νομοθετικά όργανα. Θα έχουν εκπροσώπους που θα υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους, που θα γνωρίζουν την κατάστασή τους και θα μπορούν να προασπίζουν τα δικαιώματά τους. Η κατάσταση ενός ατόμου με αναπηρία δεν μπορεί να αγνοείται στην πολιτική σκηνή. Και σταδιακά, χάρη και στις τεχνολογικές εξελίξεις, θα πρέπει επιτέλους η κοινωνία να συνειδητοποιήσει την ανάγκη να βελτιώσει την κατάσταση για τα άτομα με αναπηρία και να λάβει υπόψη τις ειδικέ τους ανάγκες. Αυτά αυτές οι ειδικέ ανάγκες των ατόμων με αναπηρία θα πρέπει να γίνουν οι πρωταρχικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αξιοποιήσουμε το δυναμικό και των ατόμων με αναπηρία και να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία. Γι' αυτό και με τις προτάσεις μας δίνουμε σάρκα και οστά στο σύνθημα του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, δηλαδή τίποτα για μας χωρίς εμάς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα να ακούσουμε την κυρία Νέστα από την Πολυνική Ένωση Υποστηρίξης των ε, Τυφλών και Κοφών. Jestem ε, osobą ε, Είμαι τυφλή και κοφή και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η ευκαιρία που δίνεται σε όλα τα άτομα με αναπηρίες να λάβουν το λόγο σήμερα και πολύ σημαντική είναι η δυνατότητα που θα έχουν τα άτομα με αναπηρίες να ψηφίσουν και για να μπορεί κανείς να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου πολύ σημαντικό είναι να έχει ε, πληροφορίες ε, και με το σύστημα Braille και κυρίως το πρόβλημα που έχουν οι κοφοί και τυφλοί είναι το, το επικοινωνιακό πρόβλημα. Θα πρέπει λοιπόν να τους εξασφαλίσουμε διερμηνία με την νοηματική γλώσσα. Θα πρέπει να υπάρχει κάποιος άνθρωπος που να μπορεί να επικοινωνήσει με τον άνθρωπο που είναι κοφός και τυφλός. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσουμε τέτοιου είδους υπηρεσίες για να διευκολύνουμε την προσβασιμότητα στα εκλογικά κέντρα των ατόμων με αναπηρία, ιδιαίτερα στην περίπτωσή μας των τυφλών και ακοφών. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμότατα. Ευχαριστώ θερμότατα όλους τους ομιλητές. Σας ευχαριστώ για την προσήλωσή σας, την αφοσίωσή σας και τις συγκεκριμένες προτάσεις σας. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους και ευχαριστώ και τους διερμηνείς που συνέβαλαν στην ευρυθμή διεξαγωγή αυτής της συζήτησης. Και εμείς ευχαριστούμε. Και τώρα να ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Ιωάννη Βαρδακαστάνη, που είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ των Ατόμων με Αναπηρία. Σας ευχαριστώ, κύριε Πουρά. Και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το τον κύριο Άνταμ τον κύριο Μάρεκ Πλούρα και την αγαπητή συνάδελφο Μωρίν Πιγκό για την ε, εξαιρετικό συντονισμό του πρώτου μέρους της εκδήλωσης. Να ευχαριστήσω επίσης όλους όσοι πήραν το λόγο. και μας έδωσαν σημαντικές πληροφορίες. Γνώση βασική που διευρύνει το πεδίο εφαρμογή τη εργασία μα. Να ευχαριστήσω επίση τους, τον αγαπητό συναδέλφο, μάλλον, τον κύριο Κλάρκ. Τον κύριο Κλάρκ ε, για το μανιφέστο με τι ευρωεκλογέ για το 2019. Με την ολοκλήρωση του πρώτου τμήματος και ελπίζουμε με την υιοθέτηση του μανιφέστο για τις ευρωεκλογέ, ξεκινάει η εκστρατεία. Και έχουμε υποχρέωση αυτή η εκστρατεία να φτάσει σε όλες τις γωνιές της Ευρώπης. Για μένα λοιπόν πιστεύω Μάλλον ε, τώρα θα περάσουμε στην επίσημη διαδικασία έγκρισης του μανιφέστο. Θα ήθελα να σας πω ότι όλα όσα μας είπατε τα σημειώσαμε. Και θα τα αξιοποιήσουμε αναλόγως. Όπως σας είπα, τώρα ξεκινάει η εκστρατεία. Επισήμως λοιπόν σας ερωτώ όπως κάνουμε και στις ε, συνεδριάσεις ε, του EDF. Είναι κανείς κατά της πρότασης όπως παρουσιάστηκε, όπως και συζητήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες με όλους τους φορείς. Μωρήν, δεν βλέπετε κανένα να ενίσταται. Αποχή, απέχει κανείς. Ως εκ τούτου συμπεραίνω ότι ομόφωνα εγκρίνεται το μανιφέστο. Πάρτε το στα χέρια σας και χρησιμοποιήσετε ως όπλο για προσβασιμότητα στις ευρωπαϊκές εκλογές. Ας φέρουμε πιο πολλά άτομα με αναπηρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως μέλη το 2019. Έχουμε το αριθματικό στοιχείο, έχουμε και το κουράγιο. Τα έχουμε όλα prove what to the right have, have banners saying right vote for all and European flagging. Thank you all, colleagues. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι, σας ευχαριστώ όλους σας. Και τώρα νομίζω ότι όλοι μας αξίζει να πάμε για μεσημεριανό. Όμως, θα πρέπει να συμπεριφερθούμε όπως ως τώρα, να τηρήσουμε τα χρονικά όρια στις 2 ε, παρα 10 όλες στην αίθουσα. Καλό μεσημέρι και στις 2 παρα 10 τα ξαναλέμε.